Chers collègues, nous allons commencer. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα αρχίσω. Παρακαλώ καθίστε. Θα προεδρεύσω εγώ σήμερα. Σας ζητώ υπομονή και κατανόηση. Πρώτη φορά προεδρεύω. Αρχίζουμε με την έγκριση του σχεδίου μέσης διάταξης. Θα ήθελε κάποιος να προτείνει προσθήκη. Όχι. Το τρίτο σημείο είναι η έγκριση των πρακτικών της συνεδρίας που έγινε στις 3 Σεπτεμβρίου 2014. Διαβάσατε νομίζω όλοι τα πρακτικά. Έχετε παρατηρήσεις, ε, θέλετε να προσθέσετε κάτι, όχι. Ε, σημείο 4. Ανακοινώσει τη Προέδρου. Πρώτη ανακοίνωση στα αγγλικά θα τα κάνω, διότι μου έστειλαν το έγγραφο στα αγγλικά. Ε, ε, μια ειδική εκπαίδευση για το gender mainstreaming στις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου θα λάβει η χώρα στις 16 Οκτωβρίου και ένα εργαστήρι στις 19 Οκτωβρίου. Ο στόχο είναι να υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και αύξηση των γνώσεων για τα ζητήματα που σχετίζονται με την ισότητα των δύο φύλων και την ενσωμάτωση τη διάσταση του φύλου στο νομοθετικό νομοπαρασκευαστικό έργο του Κοινοβουλίου. Ε, οι πολιτικοί σύμβουλοι αλλά και οι βοηθοί των βουλευτών μπορούν να συμμετάσχουν. Δεύτερη ανακοίνωση. Οι υποψήφοι ε, μάλλον ε, η Ραλά ε, Μαλάλα και η Κάισα Μασαϊτή που κέρδισαν τον Νόμπελ Ειρήνης. Η Μαλάλα θυμάστε το 2013 πήρε το βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία της σκέψης και προβάλλει το ρόλο των γυναικών και των παιδιών στον κόσμο και κυρίως το θέμα της εκπαίδευσης των γυναικών και κοριτσιών που θα είναι το βασικό θέμα στη Διεθνή ημέρα των γυναικών το 2015. Ε, μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο ζήτημα. Ε, οι συντονιστέ, οι συνεδρίε των συντονιστών στι 13 Οκτωβρίου δεν μπόρεσα να παρευρεθώ ούτε και κανένα άλλο αντιπρόεδρο ή κάποιο από το Προεδρείο. Θα ε, σας διαβιβάσουμε γραπτός τα αποτελέσματα της ε, σύσκεψης των συντονιστών και θα το συζητήσουμε ε, την επόμενη φορά. Μπορούμε τώρα να πάμε στο σημείο 6, πρόεδρος που έχει σημειωθεί ως προς την ισότητα των δύο φίλων το 2013, ο κύριος Ταραμπέλα είναι ο εισηγητής μας. Ξεκινήσαμε την περασμένη φορά την ε, συζήτηση, θα τη συνεχίσουμε. Έχουμε μια δημόσια ακρόαση. Σα υπενθυμίζω ότι κάθε χρόνο ε, γκρίνεται μια ετήσια έκθεση για την πρόοδο που σημειώνεται ω προ την πρόθεση ισότητα των δύο φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 24 Σεπτεμβρίου έγινε μια πρώτη ανταλλαγή. Ο κύριο Ταραμπέλα μα παρουσίασε τα βασικά ζητήματα που θα πραγματευτεί στην έκθεσή του. Σήμερα καλωσορίζουμε και την κυρία Ζενοβέβα Τίσεβα που είναι στα δεξιά μου και την κυρία Κλόντια Μέν στα αριστερά μου είναι οι δύο ε, εμπειρογνώμονες που θα μας παρουσιάσουν ε, τα απορίσματά τους ε, για τα φαινόμενα βίας κατά των γυναικών και την ενσωμάτωση της διάστασης των φύλων. Η κυρία Μένη είναι γραμματέας της Ευρωπαϊκής Νομοσπονδίας Συνδικάτων και η κυρία Τζενοβέφα Τίσεβα είναι από το Βουλγαρικό Ερευνητικό Ίδρυμα για την Ισότητα των Φύλων. Κύριο Σταραμπέλ. Ευχαριστώ, πολύ. Δεν έχω να προσθέσω πολλά σε αυτά που είπατε. Είχα κάνει και κάποια σχόλια στο τις προηγούμενες μέρες για την έκθεση αυτή. Το Κοινοβούλιο ήθελε να έχει μια έκθεση που θα ασχολιόταν με την ε, πρόοδο αλλά και τα προβλήματα που υπάρχουν για τα θέματα ισότητας. Εγώ ήθελα να σταθώ, όπως θα θυμάστε, σε τρία-τέσσερα κεφάλαια που θεωρώ σημαντικά. Βία, κατά των γυναικών, gender gap, ε, η εξέλιξη της βίας μέσω και των κοινωνικών ε, δικτύων και σωματική βία, όπως ε, συχνά σκεφτόμαστε, αλλά ταυτόχρονα κάτι λιγότερο σύνηθες, ψυχολογική βία, παρενόχληση που γίνεται έναντι εφήβων κυρίως, είτε μεταξύ τους ή με, νέες, με τις νέες τεχνικές των κοινωνικών δικτύων που δεν μπορούμε να γνωρίσουμε άδεια μητρότητα που έχει προβλήματα εδώ και αρκετά χρόνια, προσπαθώντα να βρούμε μια λύση, ένα συμβαστικό κείμενο στο Κοινοβούλιο μεταξύ μα καταρχά. Υπάρχει μια θέση που έχει καθυστερήσει κάπως, αλλά αν υπάρξει συμβιβασμητική λύση στο σημείο αυτό, ίσως να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μια λύση που θα συνιστά ούτως ή άλλως μία πρόοδο, μία υπεραξία για τις ε, γυναίκες της Ευρώπης. Δεν ξεχνώ επικουρικά την σημασία της άδειας πατρότητας, την ανάγκη να αναδειχθεί ο ρόλος του πατέρα από τη γέννηση του παιδιού, να κάνω και μία διαφήμιση για τους πράσινους. Ε, fathers are parents too είχαν πει οι πράσινοι. ο αντίκτυπος της κρίσης, ε, οι προκλήσεις της πολιτικής, των πολιτικών ανάκαμψης, διότι η κρίση μπορεί να αντιμετωπίζεται με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με το φύλλο. Και ως, το, ως πως το πώς παρουσιάζεται η κρίση, αλλά και το πώς βιώνεται από τον πληθυσμό. Οι γυναίκες συχνά είναι εντονότερα θύματα της κρίσης και έμφαση στην πολιτική ανάκαψη. Αλλά και εδώ δεν θα πρέπει να αφήσουμε τις γυναίκες ε, στο περιθώριο της οικονομικής ανάκαμψης. Θα μιλήσω και για το φορολογικό σύστημα που συχνά πλήττει τις γυναίκες υποχρεώνοντάς τις να μην δουλεύουν ε, με πλήρη απασχόληση δεν θα μείνω πολύ στο θέμα αυτό, θα φροντίσω ωστόσο μέσω των κρατικών μηχανισμών της φορολογικής πολιτικής ιδιαίτερα να μην υπάρξει διάκριση έναντι των γυναικών. Η πρόσβαση στην αντισύλληψη και την άμβλωση ε, είναι ένα θέμα για το οποίο θα μιλήσω, είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα, δικαίωμα και αποτελεί τμήμα ενός κεφαλαίου για μένα, αλλά και η συνδιαλλαγή ιδιωτική και επαγγελματική ζωή. Σήμερα θα σταθούμε ωστόσο σε δύο ζητήματα. Βία ε, είναι ένα σημαντικό φαινόμενο, διαδεδομένο φαινόμενο, είτε μιλάμε για τη σωματική είτε για την ψυχολογική βία. Πολιτικές ε, οι πολιτικές αλλάζουν. α πούμε, δείτε το παράδειγμα της Ισπανίας. Πριν από 10 χρόνια ήταν πολύ καλύτερη, τώρα πέρασε η κρίση και άλλαξε ολόκληρη η στάση ε, και οι δυνατότητε της πολιτείας. Αυτό που είναι ανησυχητικό σήμερα είναι και η βία προς νέους, προς νέες και μεταξύ νέων. Και το gender mainstreaming στις ε, κρατικές πολιτικές θα πρέπει σε άλλες επιτροπές, όχι μόνο τη δική μας, να έχουμε το ρεφλέξ να σκεφτόμαστε. Όταν λαμβάνουμε μια ενδιαφέρουσα για τον πολίτη απόφαση, ας προσπαθήσουμε να θυμόμαστε πάντα ότι μπορεί να έχει διαφοροποιημένη επίπτωση ανάλογα με το φύλλο των ανθρώπων. Αυτό είναι κάτι νομίζω που θα πρέπει να δούμε. Τώρα είμαστε εδώ για να ακούσουμε τις εμπειρογνώμονές μας και να έχουμε μια συζήτηση. Ευχαριστώ. Η κυρία Τίσεβα, Διευθύντρια της Βουλγαρικής Υπηρεσίας Έρευνας για την Ισότητα. Ε, η κυρία Τίσεβα πρέπει να φύγει αμέσω μετά την ε, παρέμβασή της, οπότε ε, αν θέλετε να θέσετε ερωτήματα τα κάνετε αμέσω μετά. Κυρία Τίσεβα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Με χαρά και τιμή παρευρίσκομαι ενώπιόν σας στην ακρόαση αυτή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή Γυναικών. Ευχαριστώ τους οργανωτές την κυρία Γκαμπριέλ δραστήρια στην μάχη κατά τις ε, βίας ενάντια στις γυναίκες. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για τις προσπάθειές σας να ξεκινήσετε συζητήσεις για τόσο λεπτά ζητήματα, τη βία κατά των γυναικών, προσπαθώντας να διαμορφώσετε μια σφαιρική πολιτική αντιμετώπισης της βίας εν γέννη. Βεβαίως πετύχαμε πρόοδο, έχει, έχουν αλλάξει τα πράγματα, θέλουμε ωστόσο μια πιο συνολική πολιτική με ένα νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που θα αντιμετωπίζει ουσιαστικά τη βία κατά των γυναικών. Ως εκπρόσωπος της κοινωνίας των πολιτών θα σταθώ σε κάποιες διαστάσεις της δράσης μας που που στηρίζονται στην νομοθεσία, την ευρωπαϊκή νομοθεσία των τελευταίων ετών. Έχω τη χαρά και την ευκαιρία να δουλέψω σε έναν τομέα που πραγματικά αγαπώ, δουλεύοντας για τις γυναίκες στην Ευρώπη, για τις γυναίκες στη Βουλγαρία. Το κάνω με χαρά αυτό. Είμαι και νομικός άλλωστε. Και ασχολούμαι με το θέμα της ισότητας των φίλων και της καταπολέμησης της βίας εις βάρος των γυναικών. Νομίζω ότι μπορούμε να, να βοηθήσουμε τις γυναίκες συγκεκριμένα και θα σας πω πώς, με κάποια παραδείγματα. Επίσης, θέλω να κάνω μια επισκόπηση της σημερινής κατάστασης αρχικά να αναφερθώ στο τι έχουμε πετύχει στον τομέα αυτό. Πιστεύουμε ότι το πλαίσιο αυτό είναι εξαιρετικό και καλή αφετηρία για την μελλοντική μας δουλειά και την επερχόμενη νομοθεσία. Για να χτυπήσουμε τη βία, να βοηθήσουμε τα θύματα, και την διακίνηση ανθρώπων. Πίστευουμε ότι ο αγώνας αυτός θα πρέπει να ενταχθεί σε έναν πολυσχηδή και πιο εκτεταμένο αγώνα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πριν υιοθετηθεί με δύση διάταξη για το 2015, μετά το 2015, τώρα δηλαδή, ε, βρισκόμαστε στη φάση υιοθέτησης μιας σειράς στόχων Πιστεύουμε ότι η ισότητα των φύλων και η καταπολέμηση της βίας πρέπει να ενταχθεί στο πλαίσιο αυτό. Και νομίζω ότι όλοι μας θα πρέπει να συμβάλλουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Άλλωστε, η αναθεώρηση της διαδικασίας του Πεκίνου συνεχίζεται. Επίσης, θα τονίσω το θέμα της υλοποίησης της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Πολύ λίγες είναι οι χώρες που έχουν κυρώσει τη σύμβαση αυτή. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό να ασκηθεί η πίεση προς τα κράτη-μέλη της Ένωσης, ζητώντας τους να υπογράψουν και να ακυρώσουν την σύμβαση αυτή να χαιρετήσω μάλιστα και τις χώρες ε, που επικύρωσαν τη σύμβαση αυτή, Μάλτα, Σουηδία και άλλες. Δεδομένης της ε, υφιστάμενης οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης στη Βουλγαρία, ε, οι γυναίκες необходимостта в οι γυναίκες έλεγα μπορεί να πέσουν θύματα του κοινωνικού αποκλεισμού. Η κύρωση λοιπόν της ε, Οσάνο Συμβάσεως αποτελεί προτεραιότητα δι' μας. Η μελέτη του ΦΡΑ, του Fundamental Rights Agency, είναι μια εξαιρετική μελέτη, μοναδική, που μας επιτρέπει να αναλάβουμε μέτρα παρακολούθησης και να δοθεί συνέχεια σε αυτά. Για να δούμε πώς οι χώρες αυτές, τι έκαναν οι χώρες αυτές. Τώρα, κάποια ευρωπαϊκά στοιχεία, δεδομένα. Η Βουλγαρία βρίσκεται περίπου στο μέσο όλων των ευρωπαϊκών ε, χωρών. Ωστόσο, οι υπηρεσίες που παρέχονται στις γυναίκες είναι περιορισμένες οικονομικά. Οι γυναίκες λοιπόν απειλούνται. Πάντω, Така че считаме, че трябва да се отчете това и България да Πάντως, αν δεν ληφθούν μέτρα, θα επιδεινωθεί η κατάσταση και θα πρέπει να παροτρινθεί η Βουλγαρία να, να λάβει αυστηρότερα μέτρα. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα πρέπει να συμπληρώνονται από στοιχεία που παίρνουμε μόνιμα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι αλλάζουν οι μορφές της βίας. Οι μεταναστευτικές ροές που προκύπτουν τα τελευταία χρόνια συνιστούν επιπρόσθετη απειλή. Δεν υπάρχουν οι για να οργανωθεί κατάρτιση ούτως ώστε να υπάρξει, να προληφθεί η βία κατά των μεταναστών γυναικών, για παράδειγμα από τη Συρία. Ε, θα ήθελα ωστόσο να σας δώσω και κάπως μια πιο αισιόδοξη νότα στην ομιλία μου. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με την κυβέρνηση. Η νομοθεσία της χώρας για την προστασία των γυναικών από την ε, οικογενειακή βία είναι ένα εξαιρετικό κείμενο που εφαρμόζεται στην πράξη και που είναι υποφελής για τις γυναίκες. Βάσει των στοιχείων που έχει συλλέξει η αστυνομία έχουν ε, εκδοθεί δι πάνω από 2.000 διαταγές προστασίας βάσει του νόμου αυτού και θέλω να υπογραμμίσω εκ νέου ότι οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις παίζουν ένα εξαιρετικά σημαντικό ρόλο για να βοηθήσουν τα θύματα να αναλάβουν τις απαραίτητες, ε, τα απαραίτητα διαβήματα ή να προχωρήσουν δικαστικά τις απαιτήσεις τους. Το 2014 ο νόμος αυτός εντάχθηκε στον κατάλογο των νόμων του World Future Council ως ένας από τους καλύτερους νόμους. Φέτος θα λάβει και βραβείο σχετικά και είμαστε περήφανοι για αυτή την εξέλιξη. Τώρα, σε ό,τι αφορά την μεταρρύθμιση του ποινικού κώδικα, δυστυχώς εκεί δεν έχουμε τόσο μεγάλη πρόοδο. Ο νέος ποινικό κώδικας δεν έχει εγκριθεί ακόμα. Το σχέδιο του ποινικού κώδικα προέβλεπε και συγκεκριμένα συμπληρωματικά μέτρα προστασίας των γυναικών από τη βία. Κάθε είδους ε, μορφή βίας κατά ε, το γυναικών. Μια άλλη ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία είναι η οργάνωση από το 2000, η διοργάνωση από το 2004 και μετά σε συνεργασία με δυτικούς εταίρους ενός Διεθνούς Ινστιτούτου για τα Δικαιώματα των Γυναικών. Αποκτήσαμε μεγάλη εμπειρία με τον τρόπο αυτό, έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα, το Ινστιτούτο εκπαιδεύει νομικούς από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη αλλά και την Ασία και την Αφρική σε θέματα βίας κατά των γυναικών υπό κάθε μορφή αναπαραγωγικά δικαιώματα και δικαιώματα στην εκπαίδευση και την εργασία. Οι νέοι νομικοί λαμβάνουν εκπαίδευση και κατάρτιση στο θέμα της πρόληψης και της ενημέρωσης. Χρησιμοποιούμε τα νομοθετικά κείμενα του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε κατατήσει καμιά εκατοστή νομικούς από 20 χώρες, τη Βουλγαρία, από τις γειτονικές χώρες, αλλά και από το Καζακστάν, το Ουσμπεκιστάν και άλλες χώρες. Имаме вече наблюдатели от там и да видим Τα μαθήματα αυτά είχαν ξεκινήσει για την κεντρική Ευρώπη, αλλά ε, έδειξε ενδιαφέρον, έδειξαν ενδιαφέρον και αφρικανικές χώρες, οπότε προσαρμόζουμε το πρόγραμμά μας και το, τη διδακτική ύλη στις, στα ειδικά χαρακτηριστικά των χωρών αυτών. Πιστεύουμε ότι θα ήταν χρήσιμο να συνεχιστούν οι πρωτοβουλίες αυτές. και με εξαιρετική πρωτοβουλία. Αυτό είναι μια φωτογραφία των μαθητών της εκπαίδευσης αυτής. Всеки път с около 20-25 души Οι διδάσκοντες είναι Ευρωπαίοι, Δυτικοευρωπαίοι, Ανατολικοευρωπαίοι, Αμερικανοί και αν σας ενδιαφέρει μπορώ να πω σε περισσότερες λεπτομέρειες για, την, για το Ινστιτούτο αυτό. Η τέταρτη φουρνιά των νομικών αποφύτησε πρόσφατα. Επίσης έχουμε θεσπίσει μια στρατηγική μια στρατηγική που θα παροτρύνει τις χώρες να οργανωθούν καλύτερα υιοθετώντα ε, ένα σωστό νομοθετικό πλαίσιο και διαμορφώνοντας μονάδες οι οποίες θα μπορούσαν να κάνουν κατάρτιση των γυναικών. Το κάναμε αυτό στη χώρα μας. Έχουμε πολλά παραδείγματα δικών και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου административния протокол към конвенцията СИДО. Ето тук два примера. Джало. Се συνεργαζόμαστε, συνεργαζόμαστε και με την Επιτροπή για τις Γυναίκες του, του ΟΗΕ, της ΕΝΤΑΟΥ, Ανέφερα νομίζω δύο δίκες που αφορούσαν τη Βουλγαρία και ήταν ε, οικογενειακή βία. Πιο σωστά ήταν δίκες προστασίας παιδιών και των μητέρων τους. Τζάλο κατά Βουλγαρίας και Μπεβάκουα κατά Βουλγαρίας. Στην πρώτη περίπτωση η κυρία Τζαλάου ήταν μια πολίτης Γαμβίας που χρειαζόταν προστασία όπως και τα παιδιά της.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 Βάσει του πρωτοκόλου αυτού, μάλλον οι γνωμοδοτήσεις του πρωτοκόλου αυτού αναγνωρίζονται. Ωστόσο, αντιμετωπίζουμε προβλήματα όταν θέλουμε να ζητήσουμε αποζημίωση για τα θύματα. Γιατί πρόκειται για συστάσεις και όχι αποφάσεις όπως είναι οι αποφάσεις του Δικαστηρίου του Στρασβούργου. Και αυτό είτε είναι αποζημίωση στις ίδιες τις γυναίκες είτε προς τα μέλη της οικογένειάς τους. Όπως σας έλεγα, η βία κατά των γυναικών, η αντιμετώπιση μάλλον της βίας κατά των γυναικών δεν είναι αρμοδιότητα της Ένωσης. Πρέπει ωστόσο το θέμα αυτό να μπει ούτως ώστε να μπορέσουν ε, να έχουμε δικαστικές περιπτώσεις ή δικαστικές υποθέσεις ενώπιον του δικαστηρίου της Ένωσης. Έχουμε περιπτώσεις θυμάτων που που ενός ε, θύματος που ξεκίνησε ε, δικαστική δίωξη ε, μετά, από έναν θάνατο που ζητά την κύρωση της σύμβασης. Ο στόχος, στόχος μας είναι να υπάρξουν δίκτυα, να υπάρξει ένα δίκτυο, να δημιουργήσουν δηλαδή μια σειρά δικτύωσης και συνεργασία μεταξύ των διάφορων δομών. Εμείς υιοθετήσαμε μία οργάνωση που αγωνίζεται για τα δικαιώματα των γυναικών. Έχουν ξεκινήσει κάποια κέντρα σε 11 πόλεις της Βουλγαρίας με στόχο την αντιμετώπιση και της οικογενειακής βίας αλλά και της βίας κατά γυναικών Ρωμά, κατά μεταναστριών ή κατά γυναικών που ανήκουν σε άλλες εθνοτικές μειονότητες, γυναικών που, είναι, που έχουν αναπηρία, κατά της εκτομής και άλλων ε, Δύο πρακτικών εις βάρος των γυναικών. Έχουμε μια στενή συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς. Έχουμε ένα κέντρο, εδώ βλέπετε το χάρτη των κέντρων ενημέρωσης. Βέβαια δεν έχουμε αρκετά χρήματα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε τέλο πάντων. βρισκόμαστε στην παραμονή μιας καμπής. Θέλουμε να θεσπίσουμε ένα ευρύ στρατηγικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και κάθε μορφής βίας, της βίας στα μέσα ενημέρωση, στην εκπαίδευση, така μας είναι να να, να υπάρξει πανευρωπαϊκά ένα σύστημα due diligence. Θέλουμε να υπάρξει επικύρωση της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, υιοθέτηση νομοθετικών εργαλείων που θα εξασφαλίσουν την συνέχεια της εφαρμογής της σύμβασης μέτρα πρόληψης και να μειώσουμε την και να αντιμετωπίσουμε τη διακίνηση γυναικών, να υπάρξουν μέτρα αποζημίωσης και πιστεύουμε ότι τα κράτη δεν είναι παρκώς υπεύθυνα όταν οι πολίτες τους είναι θύματα παραβίασης των δικαιωμάτων τους. Είναι επίσης αναγκαίο να υπάρξει, να δοθεί συνέχεια και να παρακολουθούν τα κονδύλια που έχουν δοθεί για την αντιμετώπιση της βίας κατά τον γεννού, γιατί πολύ συχνά οι πόροι αυτοί δεν χρησιμοποιούνται επαρκώς. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Ερωτήσεις τώρα, μία ή περισσότερες προς την κυρία Τίσεβα. Όποιος θέλει να θέσει ερώτηση τώρα, να την κάνει. Can I ask, I apologize Επιτρέψτε μου να ρωτήσω, μπορεί να ε, το έχασα διότι άργησα κάποια λεφτά, αλλά μπορείτε να μου πείτε πώς χρηματοδοτήσετε. Χρηματοδοτήσετε από κυβέρνηση, από ίδρυμα. По отношение на нашата организация, Български център за джендър изследвания, ние съществуваме. Ένα κέντρο μελετών ε, το κέντρο μελετών υπάρχει εδώ και 15 χρόνια και χρηματοδοτείται από ε, δωρητές, από τον ιδιωτικό τομέα. Από το Ίδρυμα της Βουδαπέστης, ε, το Ίδρυμα της Ομάδας της Γενέβης. Διαρκώς αναζητούμε άλλες δυνατότητες χρηματοδότησης. Βλέπετε ότι έχουμε πάρα πολλές δραστηριότητες. και χρειαζόμαστε ιδιωτικά κονδύλια βεβαίως λαμβάνουμε και από το Υπουργείο Δικαιοσύνη κάποια χρήματα καθώς και από ενώσεις που ανα... έχουν αντίστοιχε δραστηριότητες ε, για την καταπολέμηση της βίας ε, κατά των γυναικών και βάσει και του νέου νόμου Ε, χρηματοδοτούνται όλα τα ιδρύματα που ε, έχουν τέτοιες δραστηριότητες. Ε, δυστυχώς δεν είναι τακτική η χρηματοδότηση. Ε, ευχαριστώ, λέει η κυρία Γκαβρέλ. Ε, την με την κυρία Τίσεβα για την παρουσίασή της. Σε δύο ερωτήσεις έχω. Από ό,τι καταλάβαμε, πιέζετε και εσείς ούτω ώστε τα κράτη-μέλη να κυρώσουν τη σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη. Τι είδου πίεση μπορεί να ασκήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με ποια προθεσμία, ποια είναι τα ζητήματα, τα βασικά ζητήματα, Πώ μπορούν να, μπορούμε να επιτύχουμε μια ε, μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των κρατών μελών. Πρέπει και εμείς ε, να πάρουμε τη σκητάλη και να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας, ούτως ώστε να έχουμε αυτά και χρήσιμα αποτελέσματα, όχι μόνο για τις γυναίκες, αλλά και για το σύνολο της κοινωνίας. Ε, επίσης, μιλάτε για τη βία και αυτό που είναι το σημαντικότερο για μένα είναι η πρόληψη και αυτό από πολύ μικρή ηλικία. Μπορείτε να μας μιλήσετε περισσότερο για το ρόλο της παιδείας, αυτά τα κλισέ που ε, τα στερεότυπα που πολύ γρήγορα μεταδίδονται στο εκπαιδευτικό σύστημα, πώς μπορούν να καταπολεμηθούν, ε, ούτως ώστε μεταγενέστερα να μην έχουν τόσο ε, βαριές επιπτώσεις. Κάτι άλλο που μου τράβηξε την προσοχή στην παρουσίασή σας είναι αυτό που είπατε για την προστασία των προσφύγων όλο και περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ήπειρος θα έρχεται αντιμέτωπη με αυτές ε, τις καταστάσεις και όχι μόνο η Βουλγαρία, η Μάλτα, η Ιταλία, οι χώρες που βρίσκονται στα σύνορα, γιατί είναι, πρόκειται για ζήτημα ενσωμάτωσης ε, των γυναικών προσφύγων στην ε, κοινωνία και ε, θα έπρεπε να εξετάσουμε διεξοδικότερα αυτό το ζήτημα εμείς ως Επιτροπή Γυναικών και να καταθέσουμε συγκεκριμένες προτάσεις συνειδητοποιούμε όλο ένα και περισσότερο ότι χρειάζεται μια ε, κοινή μεταναστευτική πολιτική και σίγουρα αντίθετα με άλλες πολιτικές ε, θα έπρεπε να προβληθεί η σημασία ε, της γυναικείας διάστασης κατά την εκπόνηση αυτού του κοινού μεταναστευτικού πλαισίου. Σας ευχαριστούμε πάντως για τις προτάσεις σας. Ευχαριστούμε θα απαντήσω σε αυτές τις δύο ερωτήσεις της κυρίας Γκαμπρέλ με τη σειρά που τις θέσατε. Για την σύμβαση της Κωνσταντινούπολης μπορεί να αποτελεί παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση προσχωρώντας τη σύμβαση. Τι συμβαίνει συχνά ότι δεν έχει κυρωθεί από πολλά κράτη-μέλη της Ένωσης αυτή τη σύμβαση αληθεύει ότι οι πρώτοι που κύρωσαν σύμβαση ήταν εκτός Ένωσης. Δύσκολα μπορούμε να πείσουμε τις ε, κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ένωσης, διότι κάποιοι ισχυρίζονται ότι δεν πρέπει να σπεύσουμε, δεν πρέπει να κυρώσουμε άμεσα την σύμβαση. Αυτό που μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσφέρει ένα ευρύτερο πλαίσιο για την καταπολέμηση της βίας που πλήττει τη γυναίκα, να ενημερώνει τα θύματα για τα δικαιώματα που έχουν, τα δικαιώματα νομικής προστασίας εάν συνέβαινε αυτό από πλευρά της Ευρωπαϊκή Ένωση ίσως θα, μπορούσε, μπορούσαμε να μεταπίσουμε την κυβέρνηση της Βουλγαρίας, σε παραδείγματος χάρη, για να κυρώσει αυτή τη σύμβαση. Εξάλλου έχουμε μια καμπάνια στο κοινοβούλιο μας για την κύρωση αυτή τη σύμβαση. Δηλαδή θα είναι ένα ε, έφορο έδαφος η Ευρωπαϊκή Ένωση για να καλλιεργήσουμε τέτοιες ε, δράσεις ευαισθητοποίησης. Χρειαζόμαστε ένα ευρύτατο δίκτυο όπου ε, θα συνεργάζονται διάφοροι οργανισμοί, διάφορες ενώσεις για να μπορέσουμε ε, να ασκήσουμε πίεση. Ε, στη συνέχεια, για το εκπαιδευτικό σύστημα, δεν μπορούμε πλέον να δεχόμαστε αυτή την κατάσταση όπου οι γυναίκε δεν γνωρίζουν καν ποια είναι τα δικαιώματά τους. Τώρα επανέρχομαι στο πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να εγγραφούν οι προσπάθειές μας. Φυσικά πρέπει να ρίξουμε το βάρος στην πρόληψη. Εάν έχουμε φτάσει στη δίκη, πάει να πει ότι έχει υποστεί ε, τη βία η γυναίκα. Θεωρούμε πως ε, θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε με πιο πρακτικό τρόπο ε, ένα ερωτηματολόγιο, παραδείγματος χάρη, ε, που θα υποβάλουμε στις ε, γυναίκες αυτές στα κέντρα υποδοχής προσφύγων. Ε, καλό θα ήταν να έχουμε ένα ενιαίο τέτοιο ερωτηματολόγιο για όλα τα κέντρα. Οι πρόσφυγες περιμένουν περισσότερα από εμάς Προεδρεύουσα. Έχουμε και πολλές ερωτήσεις. Θα προχωρήσουμε. Μπιλμπάο Μπαραντίτσα και στη συνέχεια θα δώσουμε στην κυρία Νέλη το λόγο. Ευχαριστώ. Και καλώς ήρθατε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσίασή σας. Θέλω να ρωτήσω ωστόσο κάτι. Με αυτή τη δουλειά που κάνετε, δεν ξέρω αν το κατάλαβα καλά, κάνετε μια δουλειά η κατά τις βίας των γυναικών. ιδίω στα πλαίσια των ΜΚΟ. Ένα από τα προβλήματα όμως σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ότι ακόμα κάποιες χώρες συνεχίζουν να πιστεύουν πως η έμφυλη βία είναι ιδιωτικό ζήτημα, όχι δημόσιο. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν ότι αν αυτή η καλή συνεργασία που αναφέρεται με τις ε, κρατικές αρχές της Βουλγαρίας έχει αποδεχθεί την ανάγκη να υπάρχουν ε, προγράμματα με συγκεκριμένο προπολογισμό για να αντιμετωπιστεί όχι μόνο η έμφυλη βία που είναι συνέπεια της ανισότητας αλλά ούτω ώστε να υπάρξει και παρέμβαση σε πολιτικές ισότητας μέσω της εκπαίδευσης με προγράμματα κατάρτισης προσωπικού των σε κάθε θεσμικό όργανο. Θα ήθελα επίσης να ξέρω αν έχετε ένα Ινστιτούτο για τη γυναίκα που σε άλλες χώρες απαιτέλεσε την βάση για την διαμόρφωση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και κατάρτισης ε, για την ε, ε, ισότητα. Συμφωνώ μαζί σας ότι το 2005 στη χώρα των Βάσκων ενσωματώ υιοθετήθηκε ένα νομοθετικό κείμενο για την ισότητα όπου η, περιλαμβανόταν ολοκληρωμένο η αντιμετώπιση της έμφυλης βίας. Ε, θέλω επίσης να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι είναι χρήσιμο σε ευρωπαϊκό επίπεδο να έχουμε ένα εγχειρίδιο καλών πρακτικών. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δώσει ένα μήνυμα για τη Βουλγαρία. Να σας πω το εξής, δεν υπάρχει νόμος για την ισότητα των φύλων. Πριστάκης παλέψαμε για κάτι τέτοιο, αλλά ποτέ δεν έφτασε σε δεύτερη ανάγνωση. Είχαμε μετάσχει πάντα στη διαδικασία αυτή Αυτός ο νόμος είναι το κλειδί του προβλήματος. Ακόμα και τώρα δεν υπάρχουν εξειδικευμένα όργανα. Υπάρχει ένα συμβουλευτικό όργανο για την ισότητα των φύλων μόνο και ένα, μια διεύθυνση στο τμήμα κοινωνικών υποθέσεων που ασχολείται εν μέρη με την ισότητα. Μεταξύ άλλων προβλημάτων όπως της διάκρισης. Ακόμα και όταν πιστεύουμε ότι τούτο δεν ανταποκρίνεται στην ε, υφιστάμενη νομοθεσία, πρέπει να σας πω ότι η Βουλγαρία δεν εφαρμόζει πλήρως την οδηγία. Το πρόβλημα συνεχίζει να υπάρχει. Υπάρχουν πάντα κάθε χρόνο προγράμματα ισότητας που γίνονται δεκτά και υιοθετούνται με, συγκεκριμένα, με συγκεκριμένη περιγραφή αλλά τα οποία γίνονται από το Υπουργείο, αλλά μέσα στο πλαίσιο εφιστάμενων προπολογισμών. Δεν υπάρχει δηλαδή ειδικό προπολογισμό για την ισότητα των δύο φύλων. Η κυρία Νόηχο. Μιλήσατε για την βία εις βάρος των γυναικών υπό διάφορες ε, μορφές. Ε, υπάρχει ε, η σωματική βία, η ψυχολογική και αυτή που συνδέεται με το σεξ. Θα ήθελα να ρωτήσω τι δυνατότητες υπάρχουν για θεραπεία των γυναικών. Η σεξουαλική βία αφήνει βαθιά σημάδια στην ψυχή και απαιτείται επαγγελματική βοήθεια επί σειρά ετών. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς έχουν τα πράγματα στη χώρα σας. да ви се Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Στην Επιτροπή Συντάμ πειρασπιστήκαμε μια νεαρή κοπέλα από την Ήπεθρο που έπεσε θύμα σεξουαλικής βίας. Ήρθε αυτή η κοπέλα από την επαρχία με τη, με τη μητέρα της συγγνώμη διότι ο ένοχος ε, δεν τιμωρήθηκε. Δεν υπάρχουν ουσιαστικά μέτρα προστασίας των θυμάτων. Τα θύματα δηλαδή πρέπει μόνα τους να κινητοποιηθούν, να κινήσουν τη διαδικασία, αλλιώς εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μετά από αυτή την ε, σεξουαλική επίθεση έγινε διπολική κοπέλα και ε, προσπαθούσε με κάποιο τρόπο να ε, αντισταθμίσει αυτή την τραυματική τραυματική εμπειρία με την απόκτηση μιας αποζημίωσης και ξεκίνησε τη δίκη η μητέρα της. Προς το παρόν δεν μπόρεσε να λάβει αποζημίωση. Ανάμεσα στα υπόλοιπα καθήκοντα μας προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα θύματα διότι χρειάζονται περίθαλψη, χρειάζονται θεραπεία, όμως ε, δυστυχώς δεν ε, υπάρχει πλήρη συνείδηση του προβλήματος και δεν υπάρχουν σίγουρα κατάλληλες θεραπείες. Ευχαριστούμε. Η κυρία Χιμένα Μπαρίο θα κάνει τελευταία ερώτηση. Sí, muchísimas gracias. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Bueno, muchísimas gracias por su, por su presentación. Y yo quería saber si... Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Ξέρετε ή τι άποψη έχετε ή τι επιπτώσεις είχε στη Βουλγαρία το θέμα των δύο οδηγιών των οποίων ήμουν εισηγήτρια με την Επιτροπή Γυναικών και την Επιτροπή ε, Δημοσίων Ελευθεριών. Η μία είναι η οδηγία για την, Ευρω... για την Ευρωπαϊκή Διαταγή Προστασίας Θυμάτων, το ΕΠΟ, European Protection Order, η άλλη είναι η οδηγία υποστήριξης των δικαιωμάτων και προστασίας των θυμάτων αδικημάτων που περιλαμβάνει ένα μεγάλο κεφάλαιο για την βία κατά των γυναικών κάθε είδους, ψυχολογική, σεξουαλική, σωματική, στην εντός της οικογένειας, εκτός της οικογένειας. Θέλω να ξέρω λοιπόν Όταν ε, οι γυναίκες έχουν ε, μια διαταγή προστασίας και ταξιδεύουν σε άλλη χώρα και προστατεύονται, ήθελα να ρωτήσω το εξή. Ε, δεν υπήρξε καμία ικανοποίηση σε μια τέτοια περίπτωση όταν δηλαδή ταξίδευε μια γυναίκα. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν στην ε, Βουλγαρία πώς εφαρμόζεται. Είστε εν τω μεταξύ η οδηγία αυτή τροποποιεί το 2015. Είστε έτοιμοι να την ενσωματώσετε. Σα ευχαριστούμε. Πολύ ενδιαφέρον σε αυτή η ερώτηση για την εναρμόνιση των οδηγιών και της κείμενης νομοθεσίας. Ε, θεσπίστηκε ένας νόμος ε, για την οικογενειακή βία και βλέπουμε ότι ο δικαστής καλείται να εφαρμόσει αυτή την νομοθεσία στη συνέχεια όταν εκδίδει αποφάσεις σε διάφορες υποθέσεις θα είναι σε θέση όμως οι δικαστικές αρχές να εφαρμόσουν τις διατάξεις της οδηγίας. Ε, ως προς την απονομή της δικαιοσύνης δεν έχουν παρατηρηθεί προβλήματα μέχρι στιγμής και άρα πιστεύουμε ότι η νέα οδηγία θα βοηθήσει πολύ τις μετανάστρες στη χώρα μας. Ε, το Έχουμε μία περίπτωση επίσης εντάλματος ε, εντολής προστασίας που έχει εκδώσει, διαταγής προστασίας που έχει εκδώσει η Πολωνία. Ε, πρέπει να μεταγραφεί στην ε, Βουλγαρία αυτή η διαταγή για να μπορέσει να εφαρμοστεί. Πιστεύω ότι χρειάζεται μια ελάχιστη εναρμόνιση, κάποια ελάχιστα πρότυπα. Σίγουρα. Αυτή η οδηγία καλύπτει τα θέματα ε, κατοχύρωση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας για την ε, διαταγή προστασίας χρειάζεται εναρμόνιση. Σας ευχαριστούμε. Τώρα θα ακούσουμε την κυρία Μένε που είναι γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας ε, Συνδικάτων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, κύριοι και κυρίες Ευρωβουλευτές, ε, κύριε Ταραπέλα, σας ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα να μοιραστώ μαζί σας κάποιες ιδέες και κάποιους προβληματισμούς ε, τη Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδίας Συνδικαλιστικών Οργανώσεων σχετικά με την ενσωμάτωση της διάσταση του φύλου στην ε, δημόσια πολιτική. Ε, καταλαβαίνετε ότι μέσα σε ένα τέταρτο δεν μπορώ να εξαντλήσω το θέμα, αλλά θα προσπαθήσω να τηρήσω το χρόνο μου και να σα δώσω κάποια κίνητρα για την περαιτέρω συζήτηση. Προτού να σας δώσω κάποιες ιδέες. Θα ήθελα να πω κάποια ε, γενικά ε, θέματα, όπως είναι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, η ευρωπαϊκή κρίση, το ευρωπαϊκό εξάμεινο, η στρατηγική για την ισότητα, τα διάφορα εργαλεία που έχουμε και θέματα για περαιτέρω προβληματισμό. Και όλα αυτά μέσα σε 15 λεπτό. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι η ενσωμάτωση της διάσταση του φύλου μπορεί πράγματι να είναι πολύ ισχυρή ιδέα. Σήμερα ε, συχνά γίνεται αντιληπτή ω κάπως ασθενή ιδέα, αλλά θα ήθελα να σας ε, πω ότι σε καθημερινή βάση πρέπει να αγωνιζόμαστε για το θέμα αυτό. Γνωρίζω ε, για τι πράγμα μιλάω. Παρ' όλα αυτά είμαστε πεπισμένοι ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου ε, είναι μια πολύ ισχυρή ιδέα και χρειάζονται κάποιες ε, προϋποθέσεις για να εφαρμοστεί με επιτυχία. Χρειάζεται μια προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω, δηλαδή η ηγεσία θα πρέπει να είναι δεσμευμένη να εφαρμόσει μια τέτοια προσέγγιση. Θα πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες ώστε ο να γνωρίζει τι πρέπει να κάνει σαφείς ε, ε, ευθύνες και ε, σαφή εργαλεία. Δεν μπορώ να σας παρουσιάσω όλα τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Αναφέρθηκε η κατάρτιση στην αρχή της ακρόασης αυτής ή ο έλεγχος ε, τη ενσωμάτωση τη διάσταση του φύλου και δεν θέλω να ξεχάσω και το θέμα του προπολογισμού, στο οποίο θα επανέλθω αργότερα και επίσης ένα πρόσφατα ε, ανεπτυγμένο εργαλείο είναι ο δείκτης ε, της ενσωμάτωση τη διάσταση του φύλου που έχει αναπτύξει το Ίδρυμα στο Βίλνιους. Επίσης είναι μια διπλή στρατηγική, σημαίνει ότι όλοι πρέπει να ε, είναι δεσμευμένη για την εφαρμογή της, ε, αλλά χρειάζονται και οι σχετικές δομές, ώστε όλα αυτά να πάνε χέρι-χέρι. Τι σημαίνουν όλα αυτά για την ε, κρίση. Και βασίζω τις, τους συλλογισμούς μου στην έκθεση που αποτελεί την βάση της σημερινής ακρόασης. Τα συμπεράσματα του εγγράφου αυτού αλλά και άλλων είναι ότι η κρίση έχει μειώσει κάποια χάσματα όσον αφορά τις μισθολογικές διαφορές ε, αλλά ελπίζω να ε, συμμερίζεστε τη θέση μου. Αυτό δεν έχει ε, συμβεί επειδή έχει βελτιωθεί η κατάσταση για τους άντρες και τις γυναίκες ε, στην Ευρώπη. Το αντίθετο ισχύει έχουν ε, δηλαδή επιδεινωθεί οι συνθήκες για τους άντρες, δηλαδή έχουμε εξίσωση προς τα κάτω. Και Έχουμε επιδείνωση των αγορών εργασίας και ε, πιο πολλές ε, ανεπίσημες μορφές εργασίας για άντρες και γυναίκες. Ε, τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε αξιολόγηση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου όσον αφορά τις πολιτικές για να αντιμετωπιστεί η κρίση. συχνά χρησιμοποιείται η δικαιολογία ότι δεν υπάρχει χρόνος, ότι πρέπει να βιαστούμε και Γι' αυτό δεν γίνεται σωστή αξιολόγηση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου. Και όπως σας είπα, τα προϋπολογιστικά μέτρα ε, επίσης ε, δεν έχουν εφαρμοστεί με τις έρευνες που έχουμε κάνει. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί το μέτρο αυτό σε σχέση με την κρίση και θα ήθελα να σας θυμίσω το πολύ ενδιαφέρον Ευρωβαρόμετρο 371 του Φεβρουαρίου του 2013. Ζήτησε το Κοινοβούλιο να ε, διεξαχθεί αυτό το ευρωβαρόμετρο, να ρωτηθούν οι Ευρωπαίοι τι γνώμη έχουν για την ισότητα των δύο φύλων κατά τη διάρκεια της ε, κρίσης. Θα ήταν ενδιαφέρον ίσως στο εγγύς μέλλον να ξαναγίνει μια τέτοια έρευνα για να διαπιστωθεί πώς ο πληθυσμός της Ευρώπης ε, βλέπει τα θέματα της κρίσης σε σχέση με θέματα ισότητας των δύο φύλων. Κατόπιν έχουμε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο που έχει αναφερθεί στην έκθεση και από τον εισηγητή θέλει να λάβει υπόψη την ιδέα αυτή και να την εξετάσει. Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες της αξιολόγησής μας, αλλά πιστεύουμε ότι η λιτότητα και οι μακροοικονομικές πολιτικές υπερισχύουν των κοινωνικών πολιτικών. Η κοινωνική διάσταση στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο λείπει. Ζητούμε κοινωνική διάσταση και διαπιστώνουμε επίσης ότι οι συστάσεις αναχώρα τα τελευταία τρία ή τέσσερα χρόνια δεν είναι ε, συνεκτικά, δεν υπάρχει ε, συνάφεια όσον αφορά τα θέματα ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου. Έχουμε την έκθεσή μας, ε, μπορώ αν θέλετε να σας στείλω την δική μας αξιολόγηση. Συνεργαζόμαστε με το ε, αρμόδιο Ινστιτούτο μας ε, και θα διαπιστώσετε ότι για την Αυστρία υπάρχει σύσταση για τη μισθολογική διαφορά ανδρών και γυναικών, αλλά οι 27 άλλες χάρες δεν έχουν λάβει σχετική σύσταση, παρότι ξέρουμε ότι υπάρχει σχετικό πρόβλημα σε όλες τις χώρες. Γιατί λοιπόν έχει λάβει η Αυστρία τέτοια σύσταση και όχι άλλες χώρες. Εμεί ω συνδικαλιστικέ οργανώσει ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για τον κοινωνικό διάλογο, ο οποίο ε, συχνά παραμελείται ε, κατά τη διάρκεια τη ε, σύνταξη των συστάσεων αναχώρα. Ζητάμε λοιπόν περισσότερο κοινωνικό διάλογο, η κοινωνική εταίροι σε θέματα αγοράς εργασίας ε, είναι ενημερωμένοι παράγοντες και θα πρέπει να συμμετέχουν σε διαβουλεύσεις των κρατών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Υπάρχουν κοινωνικοί δείχτες, υπάρχει ο κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων, δεν είναι ε, δεσμευτικός νομικά, αλλά θα πρέπει να ενσωματωθεί και εδώ η διάσταση του φύλου και ε, Έχουμε τώρα τον ε, νέο διορισμένο επίτροπο που έχει ζητήσει αξιολόγηση του κοινωνικού αντικτύπου, κάτι που έχουν ζητήσει διάφορες με κυβερνητικές οργανώσεις και άλλοι παράγοντες ε, και μπορεί αυτό να αποτελέσει δρόμο για να εξετάσουμε ε, το θέμα της ενσωμάτωσης της διάστασης του, του φύλου. Επίσης γνωρίζετε όλοι ότι έχουμε στρατηγική ισότητα και ελπίζουμε ότι θα έχουμε μια νέα τέτοια στρατηγική και ότι θα γίνει σχετική διαβούλευση. Επίσης γνωρίζουμε ότι γίνεται συζήτηση σχετικά με την ομοθετική κόποση τη λεγόμενη. Και θα ήθελα να σας θυμίσω η διαδικασία REFIT και παρότι κατά διάρκεια αυτή τη θητεία δεν θα υπάρχουν πολλέ δυνατότητες να εφαρμοστεί νέα νομοθεσία, υπάρχει παρόλα αυτά μακρύ κατάλογος θεμάτων ε, που εφαρμόστηκαν στην ε, προηγούμενη θητεία. Έχουμε την προστασία της ε, μητρότητας, έχουμε την γονική άδεια, την ισορροπημένη σύνθεση των διοικητικών συμβουλίων των εταιριών και η Επιτροπή Μάλλον, συγγνώμη, υπάρχουν συστάσει για τη μυθολογική διαφορά ανδρών γυναικών, οι οποίε όμω είναι λιγότερο δεσμευτικέ από αυτέ ε, τι ε, συστάσει αναχώρα και πιστεύουμε ότι υπάρχει ανισορροπία ανάμεσα σε συστάσεις οι οποίες δεν είναι ενσωματωμένες στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Επίσης υπάρχει ε, το ανοιχτό ερώτημα των άλλων μορφών άδειας για τη φροντίδα μελών της οικογενείας κλπ. Υπό το φως της ε, δημογραφικής εξέλιξης θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό επιγόντως σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο. Και τέλος έχουμε την ε, σεξουαλική βία. Έχω βάλει εδώ ερωτηματικό, δεν είμαι τόσο αισιόδοξη όσο η προηγούμενη ομιλήτρια, κρίμα που έφυγε, διότι είπε ότι υπάρχει ένα εξαιρετικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εμείς πιστεύουμε ότι παρά τις ε, εργασίες που έχουν γίνει τα τελευταία 4-5 χρόνια, Γνωρίζουμε τι ακόμα απομένει να γίνει, έχουμε στοιχεία, αλλά ε, λείπει το πλαίσιο. Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε πάνω σε τέτοιο θέμα. Θα ήθελα να αναφέρω ότι το Διεθνές Γραφείο Εργασίας ε, εκπονεί τώρα μια σύμβαση για τη σεξουαλική βία και θα συζητήσουμε το θέμα αυτό στην αρμόδια επιτροπή μας την επόμενη εβδομάδα. Πώς θα μπορέσουμε δηλαδή να στηρίξουμε τις εργασίες αυτές του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας πάνω στη σεξουαλική βία. Υπάρχουν και άλλα εργαλεία και μέσα. Όπως σας είπα δεν είναι εξαντλητικός ο κατάλογος αυτός. Ε, απλά παρουσιάζω κάποιες ιδέες που είχα κατά την προετοιμασία της σημερινής ακρόασης. Είναι θέματα που μπορούμε να δούμε σε σχέση με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου. Γιατί να μην εξετάσουμε λοιπόν ε, την εγγύηση των ε, νέων κατά την εφαρμογή της, να δούμε δηλαδή τι συνέπειες έχει για νέους και νέες. Από ό,τι γνωρίζω δεν έχει εξεταστεί αυτό μέχρι τώρα. Θα πρέπει να εξετάσουμε όμως πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε την ε, εγγύηση των νέων και επίσης το πακέτο κοινωνικών επενδύσεων. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η προσέγγιση αυτή και έχει αναφερθεί επανειλημμένα η χρηματοδότηση προγραμμάτων και η συγχρηματοδότηση, κάτι που επίσης αναφέρεται στην έκθεση. Υπάρχει σαφή δέσμευση, αλλά είναι σημαντικά τα χρήματα και θα πρέπει να δούμε πώς χρησιμοποιούνται και υπό το φως της ενσωμάτωσης ε, της διάστασης του φύλου και των άλλων δραστηριοτήτων ε, ευαισθητοποίησης. Ε, όπως σας είπα λοιπόν ο κατάλογος αυτός δεν είναι εξαντλητικός, είναι απλά κάποιες ιδέες που μου ήρθαν κατά την προετοιμασία της σημερινής ακρόασης. Και επίσης έχουμε κάποια θέματα για περαιτέρω προβληματισμό κατά την προετοιμασία μιας νέας στρατηγικής για την ισότητα των δύο φύλων, τον ρόλο των ανδρών ε, έχει εξεταστεί ε, σε ένα βαθμό, όχι όμως ε, επαρκώς. Θα πρέπει να εξετάσουμε τα στερεότυπα που υπάρχουν στην εποχή μας, διότι βλέπουμε ότι επανερχόμαστε στους παραδοσιακούς ρόλους και θα πρέπει να εξετάσουμε πάλι τα στερεότυπα. Επίσης ε, θα μπορούσα να κάνω λίγη διαφήμιση, όχι για μένα ε, ή την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, αλλά την ε, Ένωση Δασκάλων σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή της Ομοσπονδίας Ευρωπαίων Δημοσιογράφων, που είναι και αυτοί οι άνθρωποι που διαμορφώνουν την πολιτική θα μπορούσαμε δηλαδή να εξετάσουμε τα στερεότυπα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υπάρχουν ε, λοιπόν ενδιαφέρουσες ιδέες ε, με τις οποίες μπορούμε να συνεισφέρουμε στην ε, συζήτηση στο πλαίσιο των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Τελευταίο σημείο είναι το χάσμα στις συντάξεις. Θα πρέπει να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, θα πρέπει να το αναπτύξουμε αυτό περαιτέρω και να εξετάσουμε δηλαδή και τη, και τη διαφορά στη σύνταξη, όχι μόνο τη μισθολογική διαφορά. Και Τέλος, ε, στην περίοδο ανάκαμψης υπάρχουν διάφοροι τομείς που φαίνεται να έχουν δυνατότητες ανάπτυξης και θα πρέπει να εξετάσουμε τους τομείς αυτούς και να δούμε τι σημαίνουν για τους ε, νέους άντρες και τις νέες γυναίκες. Να αναφερθώ στα επαγγέλματα STEM, δηλαδή επιστήμη, τεχνολογία, επιστήμες μηχανικών και μαθηματικά. Ε, έχουμε τις λεγόμενες λευκές θέσεις εργασίες, και τις πράσινες θέσεις εργασίας. Σε όλους αυτούς τους τομείς υπάρχει η διάσταση των φύλων, την οποία θα πρέπει να εξετάσουμε και χρειαζόμαστε συλλογική δράση. Θα ήθελα να σας πω ότι είμαστε στο πλευρό σας ε, για οποιασδήποτε δράση σας ε, στην μελλοντική θητεία. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε στενά, όπως άλλωστε κάναμε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε που δεν υπερβήκατε και το χρόνο που σας αναλογούσε. Ας ακούσουμε τις ερωτήσεις τώρα. Okay, um... Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή. Βρίσκω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα παρότι απλά επισημάνατε κάποια θέματα πάνω στα οποία θα πρέπει να εργαστούμε. Βρήκα πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε για την εγγύηση των νέων νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στους νέους και στις νέες. Θα πρέπει δηλαδή να εξετάσουμε και τη συνολική πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, διότι δεν νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα αρκετά δεδομένα και στοιχεία. Έχω όμως δύο άλλες ερωτήσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με τη διαφορά στις συντάξεις ανδρών γυναικών είναι ένα θέμα που θίξαμε ε, κατά τη διάρκεια και της ακρόασης με την Μαριάννα Τάισεν, ε, διότι αν εξετάσει κανείς τη λευκή βίβλο της Κομισιόν από τη μία και από την άλλη τις συστάσεις αναχώρα που συχνά ε, δίδονται, θα διαπιστώσει κανείς σημαντική διαφορά όσον αφορά τις συστάσεις δηλαδή για την αντιμετώπιση της διαφοράς της συντάξης. Σύμφωνα με την ε, στρατηγική Ευρώπη 2020 θα πρέπει να αυξηθεί το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών. Είναι σημαντικός ο στόχος αυτός. Θα ήθελα να ρωτήσω όμως εάν πιστεύετε ότι υπάρχει ανάγκη για δράση και από την Κομισιόν και από το Κοινοβούλιο σε κάποιους ε, τομείς. Και επίσης αναφερθήκατε στην εκπροσώπηση των γυναικών στις συνδικαλιστικές οργανώσεις. παρότι στην έκθεση νομίζω λέει ότι το 45% των μελών της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδικαλιστικών Οργανώσεων ε, είναι γυναίκες, ε, είναι, αποτελούν εξαίρεση οι γυναίκες που εκπροσωπούν τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Τι κάνετε λοιπόν εντός του κινήματός σας, θα ήθελα πολύ να ξέρω. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή. Ε, θα χρειαζόμουν χρόνο για να πω σε λεπτομέρειες, αλλά ναι, πράγματι, ε, η διαφορά στις συντάξεις ε, και οι συστάσεις αναχώρα. Υπάρχει πράγματι ασυνέπεια ανάμεσα στα συμπέρασματα της πρώτης έκθεσης ε, και ε, δεν αναφέρεται το θέμα αυτό και στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Εντό τη Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων αρχίσαμε να το συζητάμε αυτό και με τι συνταξιδοτικέ οργανώσει μα το θέμα είναι πώς μπορεί κανείς να αντισταθμίσει ε, σε βάθος χρόνου την ε, διαφορά ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες ε, στην αγορά εργασίας. Γυναίκες στην ηλικία μου όταν βρίσκονται κοντά στην ηλικία συνταξιδότησης ή όταν παίρνουν σύνταξη έχουν συχνά άδειες ή γυναίκες ε, που ε, έχουν ε, άδειε διαρκείας και δεν συνεισφέρουν στο συνταξιοδοτικό σύστημα αντιμετωπίζουν προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να εξετάσουμε αντισταθμιστικά μέτρα. Αυτό όμω μπορεί να αφορά μόνο τι ε, συντάξει του πρώτου πυλώνα, δεν μπορεί να ε, αφορά του άλλου πυλώνε ε, ή τι ιδιωτικέ συντάξει. Αυτή λοιπόν η ανακατανομή μπορεί να γίνει μόνο εντό του πρώτου πυλώνα. Αυτές είναι οι πρώτες σκέψεις μας. Θέλουμε όμως να συζητήσουμε τη συζήτηση πάνω στο θέμα αυτό. Και όπως ε, σας είπα, πολύ ευχαρίστως ε, προσβλέπω στην ε, καλή συνεργασία με το Κοινοβούλιο πάνω στο θέμα αυτό. Δεν πρέπει να εξετάσουμε δηλαδή μόνο την απασχόληση, πρέπει να εξετάσουμε και άλλους τρόπους αντιστάθμισης. Και όσον αφορά το 45% των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και το την απουσία σε γενικά στην εκπροσώπηση. Είναι ένα θέμα το οποίο εξετάζουμε. Ε, η εκπροσώπηση των γυναικών ε, παραμένει σταθερή ε, εντός του συνδικαλιστικού κινήματος, ενώ η ενώ το ποσοστό των αντρών μειώθηκε κατά διάρκεια της κρίσης ε, λόγω απώλειας θέσεων εργασίας. Ε, θα πρέπει να βελτιωθεί η εκπροσώπηση. Έχουμε κάποιες διατάξεις που αφορούν την ΕΤΟΥΚ, την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία και άλλες οργανώσεις, ε, αλλά διαπιστώνουμε ότι οι υψηλέ θέσεις, γενική γραμματείς, πρόεδροι κτλ. είναι κυρίως άντρες. Στην δεύτερη ή τρίτη σειρά έχουμε πιο ισορροπημένη εκπροσώπηση που είναι η ε, επικεφαλής ε, των διαφόρων τομέων, ε, τμήματων κλπ. Η ΕΤΙΚ έχει πολύ λίγη δυνατότητα να επηρεάσει την κατάσταση αυτή. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση. Θέλω να να σχολιάσω την έκθεση Ταραμπέλα και να υποβάλω κάποιες προτάσεις και θέλω την άποψή σας. Οι ώρες εργασίας ανά την Ευρώπη διευρύνονται. Σε βράδια, Κυριακές, ε, αργίες. Η οικονομική κρίση κατέστησε εντονότερη το πρόβλημα αυτό. Στις υπηρεσίες δε όπου οι γυναίκες ε, είναι η πλειοψηφία και υποφέρουν περισσότερο. Γι' αυτό η έκθεση Ταραμπέλα, κατά την άποψή μου, πρέπει να περιλάβει την ανάλυση της υφιστάμενης νομοθεσίας και συστάσεις για το πώς θα συμβιαλλαγεί η εργασία με την ανάπαυση, ιδίως στις Κυριακές. Η έκθεση αναφέρεται επίσης και στα αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών, το βάζοντας το δικαίωμα στην ε, ε, άμβλωση μπροστά από το δικαίωμα στη ζωή. Η αναπαραγωγική υγεία είναι και, παραμέ... και πρέπει να παραμείνει αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ε, το να επιμένουμε σε τέτοια θέματα στην έκθεση σημαίνει ότι δεν θα έχει υποστήριξη και εν τέλει θα κοστίσει χρόνο και χρήμα χωρίς αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. καυτό θέμα η ώρα εργασία. Είναι δύσκολο από πλευρά ε, ε, συνδικάτων να μιλήσουμε για το θέμα αυτό, γιατί την περασμένη άνοιξη δεν καταφέρουμε να συμφωνήσουμε για ένα νέο πλαίσιο για τις ώρες εργασία, εβδομάδα, εβδομάδα και μήνα. Περιμένουμε τις μελέτες της σε εθνικό επίπεδο στον τομέα της υγείας ιδίας ε, για τις ε, υπερβολικά πολλές ώρες εργασίας στον τομέα της υγείας. Φοβόμαστε ωστόσο ότι τα κράτη-μέλη θέλουν επέκταση, δεν θέλουν να καλύψουν τις περιπτώσεις που είσαι ε, σε εφημερία και σε η οδηγία αυτή προβλέπεται να προχωρήσει την Άνοιξη. Περιμένουμε να δούμε τι θα περιέχει. Το ενδιαφέρον ήταν ότι στις διαπραγματεύσεις που είχαμε μεταξύ συνδικάτων και εργοδοτών υπήρχε μια αμοιβαία κατανόηση στο ότι στις πολιτικές συνδιαλλαγής οικογενειακής και επαγγελματική ζωής πρέπει να δείχνουμε μεγαλύτερη ευελιξία όχι μόνο προς όφελος των εργοδοτών αλλά και των ε, υπαλλήλων που έχουν καθημερινές ή εβδομαδιαίες ανάγκες που πρέπει να καλύψουν, ας πούμε επίγονται οικογενειακά ζητήματα. Αυτό είναι κοινή εντύπωση αλλά δεν καλύπτει, δεν είναι αρκετό για να αντιμετωπίσουμε συνολικά το θέμα των, ε, του χρόνου εργασίας που είναι ένα από τα πιο δύσκολα που υπάρχουν. Ευχαριστώ. Η, κυρία Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστούμε κυρία Μαν για την ε, παρουσίαση που κάνατε. Κατά πάσα πιθανότητα θα μπορούσα να υποστηρίξω τις περισσότερες συστάσεις σας, αλλά ταυτόχρονα να είμαι λίγο επικριτική, μάλλον να ζητήσω αυτοκριτική από τις πλευρά των συνδικάτων, διότι είπατε ήδη ότι η εκπροσώπηση των γυναικών στην ηγεσία των ε, συνδικαλιστικών οργανώσεων θα μπορούσε να βελτιωθεί. Λοιπόν, ε, οι συνδικαλιστικέ οργανώσει δεν βοήθησαν πάντοτε τον αγώνα των γυναικών, διότι αντιστέκεστε στη μεταρρύθμιση τη αγορά εργασία. Εκπροσωπούν ε, τα ε, συνδικάτα αυτού που έχουν δουλειά. Ωραία, εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Αυτό δουλειά σα είναι. Εξορισμού προστατεύεται αυτού που είναι ήδη μέσα. Εις βάρος των απ' πολλές φορές. Οι νέοι, οι γυναίκες, οι μετανάστες που είναι απ' έξω παρεμποδίζονται από τη δική σας δράση. Για να δούμε στη χώρα μου τι συμβαίνει. Ε, πολλοί έχουν βρει δουλειά ως ανεξάρτητοι επαγγελματίες. Ε, πολύ καλά εργάζονται στο σπίτι τους, έχουν φτιάξει μια δική τους μικρή επιχείρηση. Ανεξάρτητοι λοιπόν, χωρίς εργαζομένους είναι εκτός του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, των εξοδοτικών ρυθμίσεων, της προστασίας από το εργατικό δίκαιο, όχι επειδή το διαλέγουν, αλλά διότι δεν μπορούν να μπουν μέσα στην αγορά εργασίας και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ε, ε, μέχρι στιγμής είχαν εξαιρετικά συντηρητικό ρόλο και ε, γι' αυτό θα ήθελα να εξετάσετε και άλλα ενδεχόμενα, άλλες πιθανές λύσεις. Σε σχέση με τις θέσεις σας τώρα για τη λιτότητα, θα έλεγα ότι εντάξει, αν αντιτάσσετε στη λιτότητα, ε, που παρενθετικά να πω ότι μικρή σχέση έχει με το θέμα της διάστασης των φύλων, τότε ωραία, τι εναλλακτική προτείνετε εσείς, διότι το να παραμείνει σε αυτό το επίπεδο το δημόσιο χρέος, το ώστε το κόστος εξυπηρέτησης του να είναι υψηλότερο από τις δαπάνες για την ε, παιδεία ή για τις κοινωνικές παροχές, δεν είναι μια βιώσιμη κατάσταση, δεν είναι ε, καλό για την κοινωνία, δεν είναι αλληλέγγυο ένα τέτοιο σύστημα. Εσείς τι προτείνετε ούτως ώστε η εξυπηρέτηση του χρέους ε, να μην μας κοστίζει τόσο πολύ όσο, περισσότερο μάλλον από τις ε, δαπάνες για την παιδεία και την κοινωνική ασφάλιση για την άμβλωση τώρα εφόσον το θέσατε, καμία σχέση με την παρουσίασή αλλά εν πάση περιπτώσει είπατε ότι είναι εθνική αρμοδιότητα ε, τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα πάλι εντάσσονται σε αυτό το πακέτο της δημόσιας πολιτικής και πρέπει να ενταχθούν μακροπρόθεσμα, ε, όπως και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα υγείας, ε, σε μια ευρωπαϊκή πολιτική υγείας. Αλλά καρ δεν μπορούμε να διαλέγουμε τι είναι εθνική αρμοδιότητα και τι όχι. Ε, μέσα στο email μου έχω απίστευτα πολλές προσκλήσεις για σεμινάρια, για διάφορες επιμέρους πτυχές του συστήματος της υγείας. Ας βάλουμε και τα σεξουαλικά και αναπορογικά δικαιώματα. Είναι απαράδεκτο σε κάποια κομμάτια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρχει πρόσβαση ε, σε ασφαλή και νόμιμη άμβλωση και σε άλλες όχι. Ε, αυτό συνιστά μεγάλη αδικία. Προεδρεύουσα, σας παρακαλώ να συντομεύετε γιατί δεν έχουμε μόνο αυτό το ζήτημα στην ημερήσια διάταξη. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία ε, Μάνε για να μας απαντήσει. Έχουμε την κυρία Κοσλόσκα, Μαρίνα, Βαλίνα α, και τον κύριο Ταραμπέλα για να κλείσει αυτή τη συζήτηση εφόσον είστε εισηγητής. Είναι κάπως δύσκολο να απαντήσω σε όλες τις παρατηρήσεις γιατί είμαστε κατά της λιτότητας. Ε, το έχω εξηγήσει σε, διάφορες, σε διάφορα έγγραφα. Δεν μπορώ να σας θυμίσω όλα όσα έχουμε εκπονήσει το τελευταίο 24 μήνο. Πιστεύουμε ότι η συλλογική λιτότητα στις 28 ε, χώρες ε, της Ευρώπης δεν βοηθούν την ζήτηση Υπάρχουν πάρα πολλοί οικονομολόγοι που στηρίζουν την ιδέα αυτή και ακόμα και ο πρόεδρος Γιούγκερ ζητά σχέδιο επενδύσεων 300 ε, δισεκατομμυρίων και χρειαζόμαστε επενδύσεις και στο ανθρώπινο δυναμικό και στις υποδομές. Διότι αυτό δημιουργεί απασχόληση, θέσεις εργασίας και πρόπτικες για το μέλλον. Εάν θέλετε, μετά πίνοντα ένα καφέ έξω, μπορώ να σας ε, εξηγήσω τις λεπτομέρειες. Έχουμε υιοθετήσει δικό μα σχέδιο επενδύσεων, 2% ε, του ΑΕΠ ζητάμε, ιδιωτικές επενδύσεις, όχι μόνο δημόσίε, για να δώσουμε επανεκκίνηση στην ε, οικονομία της Ευρώπης έχουμε περισσότερες επισφαλείς θέσεις εργασίας, περισσότερες ε, ανεπίσημες μορφές εργασίας. Θέλουμε πλήρη απασχόληση και μερική απασχόληση με κοινωνική προστασία όμως και θέλουμε να καταπολεμήσουμε όλα τα παραθυράκια και τις ασυνέπειες που υπάρχουν στον εργασιακό νόμο. Υπάρχουν πάρα πολλές δημοσιεύσεις, ε, δεν μπορώ να σας δώσω πολλές λεπτομέρειες αλλά κάθε αυτοαπασχολούμενος ε, στην Ευρώπη είναι ε, ευπρόσδεκτος να συμμετάσχει στο συνδικαλιστικό κείμενο. Υπάρχει χώρος και για τέτοιες μορφές απασχόλησης. Ε, ακόμα και εσείς μπορείτε να γίνετε μέλη μιας συνδικαλιστικής οργάνωσης αν θέλετε. Δεν είμαστε ε, λέσχοι που αποκλείει το, τον κόσμο απ' έξω. Όσο περισσότεροι συμμετάσχουν τόσο το καλύτερο. Έχουμε λοιπόν διάφορες ομάδες, δεν μπορώ να σας αναφέρω όλες τις δομές που έχουμε σε όλη την Ευρώπη, αλλά υπάρχουν ε, και ε, ομάδες ε, ανέργων που μπορούν να συζητήσουν τα προβλήματά τους. Θέλουμε λοιπόν κοινωνική προστασία για όλους, είναι ανθρώπινο δικαίωμα αυτό, δεν είναι αποκλειστικό δικαίωμα κάποιων ομάδων του πληθυσμού. και λέμε ότι η εργασιακή σύνταξη θα πρέπει να είναι συμπληρωματική της σύνταξης του πρώτου πυλώνα. Είναι πολύ δύσκολο να μπω σε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά ναι, αν πιστεύετε ότι είμαστε ε, συντηρητική. Αυτό το άκουσα πρώτη φορά πριν 20 χρόνια όταν εργαζόμουν ε, στην Γερμανία. Μας λέγανε ότι ε, οι συνδικαλιστικέ οργανώσει είναι οι δεινόσαυροι του 21ου αιώνα. Εγώ πάντω εμένω στι θέσει μου, στι αξίες μου και δεν χρειάζεται κάθε πέντε χρόνια να αλλάζω τη γνώμη μου. Ναι, είμαι συντηρητική. Ε, θα περάσουμε στην επόμενη ερώτηση, κυρία Κοσλόφσκα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ ε, για τις παρουσιάσεις. Ε, νομίζω ότι όλοι όσοι υπερασπίζονται τα δικαιώματα των γυναικών έχουν ένα πολύ δυνατό σύμμαχο στα, στις συνδικαλιστικές οργανώσεις και είστε και ένας βασικός νομιλητής στο διάλογο που έχουμε με τις κυβερνήσεις. Ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχει ομοιομορφία ως προς τη θέση των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Παραδείγματο χάρη στην Πολωνία, ε, οι ενώσεις και τα λόμπι των γυναικών, μεταξύ άλλων, ε, ζητούν ευέλικτα ωράρια εργασίας. Είναι βασική η αξίωσή τους και γι' αυτό ζητούν κύρωση της Σύμβασης Κωνσταντινούπολης. Τα λόμπι των γυναικών στην Πολωνία ζητούν εφαρμογή της οδηγίας, την εφαρμογή της οδηγίας για τις ποσοστώσεις ε, ε, των γυναικών στις επιχειρήσεις και ε, από πλευράς των συνδικαλιστικών οργανώσεων όμως προβλήθη αντίσταση κατά των ευέλικτων ωραρίων εργασίας, κάτι που θα διευκόλυνε πολύ τις γυναίκες στην Πολωνία. Δεν ε, συμμετείχαν επίσης συνδικαλιστικέ οργανώσει στη συζητήσει για την κύρωση τη σύμβαση Κωνσταντινούπολης. Οι... Στις ε, επιχειρήσεις είναι σχεδόν αποκλειστικά αντρική στελέχωση, κυρίω όταν μιλάμε για τα διοικητικά συμβούλια και θα ήθελα να σα ρωτήσω, υπάρχει ελπίδα ε, με καθολικό και πάγιο τρόπο μπορούμε να ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα υπερασπίζονται τελικά τα δικαιώματα των γυναικών τα συνδικάτα. Another Και άλλη δύσκολη ερώτηση. Δεν ξέρω πώς είναι η κατάσταση στην Πολωνία. Ξέρω πώς είναι οι συζητήσεις για τα συνταξιοδοτικά. Δεν ξέρω τι γίνεται με τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Ξέρω ότι οι συνάδελφοι του Πολωνικού, της Πολωνικής Ένωσης Συνδικάτων ε, πιέζεται από την κυβέρνηση για ευέλικτη αγορά εργασία γενικότερα και για τις ελευέλικτε όρες εργασίε. Υπάρχει πάντως μεγάλη αντιπαράθεση μεταξύ των συνδικάτων και της τωρινή κυβέρνησης για τα θέματα της ευελικτοποίησης. Δεν μπορώ να σας πω γιατί. Τώρα, οι ποσοστώσει. Η ETUC οθέτησε μια κοινή δήλωση. Συμφώνησαν οι Πολωνοί. Μα άρεσε η έκθεση του ΕΚ και η πρωτοβουλία τη κυρία Ρέντινγκ και η νέα οδηγία και εγώ είχα μετάσχει στον σχεδιασμό της νέα αυτή οδηγίας. Παρότι πρέπει να σα πω ότι οι εκτελεστικοί διευθυντέ τη επιχειρήση δεν είναι ε, μεγάλο κομμάτι των, ε, του συνδικάτου μας. Η ερώτηση που θέταμε συχνά ήταν τι σας νοιάζει η ιστορία με τους ε, ε εκτελεστικούς διευθυντές. Υπάρχουν άλλοι εργαζόμενοι που έχουν πολύ περισσότερη ανάγκη. Αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς υιοθετήσαμε την πρόταση αυτή και την υποστηρίζουμε την οδηγία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η μόνη, το μόνο συνδικάτο που ρητά δήλωσε ότι δεν το υποστηρίζει είναι το συνδικάτο της Λετωνίας. Νομίζω ότι και στην Πολωνία βέβαια υπάρχουν κάποιες επικρίσεις. κυρία Ρένα. Θέλω να επανέλθω στα στερεότυπα στην παιδεία. Πριν από αυτό ωστόσο θέλω να πω ότι ανήκω στους συντηρητικού ε, που ανέφερε η τους συντηρητικούς που υποστηρίζουν τα κοινωνικά δικαιώματα. Αν αυτό είναι ο ορισμός του συντηρητικού, είμαι συντηρητική και περήφανη γι' αυτό. Να μιλήσω λοιπόν για τα στερεότυπα. Είπατε ότι υπάρχουν δύο μεγάλη, μεγάλα σημεία όπου τα στερεότυπα υπάρχουν. Εκπαίδευση, τύπος. Έχει γίνει και σχετική δουλειά. Θα μιλήσω για την εκπαίδευση ιδίως. Καταλαβαίνουμε ότι από τα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσης των παιδιών, ο 80% των, δασκάλων είναι γυναίκες και πάνω από 80% γυναίκες που ήταν και αυτές οι εισαγωγικά θύματα ενός στερεότυπου. Συχνά στράφηκαν, υποχρεώθηκαν να στραφούν στην, ε, στον εκπαιδευτικό χώρο γιατί υπέστησαν το στερεότυπο που έλεγε οι γυναίκες πάνε στα κοινωνικά, οι άντρες πάνε στην επιστήμη. Πρέπει να υπερβούμε το στερεότυπο αυτό. Πώς είναι λοιπόν ο ρόλος των συνδικάτων μέσα στην Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών για να αλλάξει η νοοτροπία και των γυναικών που ήταν θύματα και το πώς η αρχική απόφαση μπορεί να δώσει ενημέρωση για την επαγγελματική επιλογή από μικρή ηλικία. Ξέρω ότι συχνά οι διδάσκοντες δεν βλέπουν πολύ με καλό μάτι την συνεργασία με τον ε, βιομηχανικό κλάδο, γιατί θεωρούν ότι βάζουμε την οικονομία στην εκπαίδευση. Πώς μπορούμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα της μείωσης των συνόρων. Ευχαριστώ. Νομίζω, ίσως όχι μακροπρόθεσμα, αλλά μεσοπρόθεσμα, θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία. Υπάρχουν ε, κάποιες ε, ενώσεις δασκάλων που είναι πιο προχωρημένες ε, στο θέμα αυτό και άλλες που θα πρέπει να το εξετάσουν το θέμα. Συμφωνώ με την ανάλυση σας ότι στα δημοτικά είναι περισσότερες δασκάλες και λιγότεροι δάσκαλοι και ήδη είναι πρόβλημα το πώς μπορούν ε, τα παιδιά σε μικρή ηλικία να μάθουν τους διάφορους ρόλους, ε, να έχουν και δασκάλους και δασκάλες και υπάρχει και το θέμα των στερεοτύπων που προβάλλουν ε, τα βιβλία και το εκπαιδευτικό υλικό. Υπάρχει και πάντα το θέμα της συνεργασίας με τον ε, βιομηχανικό τομέα και το πώς μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα το εποπτικό υλικό στα σχολεία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Δασκάλων έχουν εξετάσει το θέμα και έχουν κάποια ενδιαφέροντα ευρήματα, τα οποία μπορώ να σας στείλω αν σας ενδιαφέρει. Σας ευχαριστούμε. Βαλίνα Sí, ε, Γεια σας. Τι άποψη θεωρείτε ότι πρέπει να έχουν δηλώσει όπως αυτές που έγιναν πριν από λίγες μέρες στην Ισπανία η πρόεδρος ε, της Ένωσης Επιχειρήσεων λέγοντας ότι ουδέποτε θα έπαιρνε γυναίκες από μεταξύ 25 και 45 ετών γιατί είναι η ηλικία της ε, γονιμότητας. Με τέτοιες τάσεις που περιλαμβάνουν διακριτική αντιμετώπιση, παράλογο, παράνομο ήδη και επιβάλλει στη γυναίκα να επιλέξει αν θα είναι μητέρα ή εργαζόμενη, τι έχουμε να κάνουμε. Και η άλλη ερώτηση είναι, αν δεν έχουμε παιδιά, ποιο πήρε πλέον τι συντάξει αύριο. Τι άποψη έχετε εσεί ω ε, συνδικαλιστέ για στάσει ε, ανθρώπων όπω η κυρία που είναι γυναίκα, επιχειρηματίας και μητέρα έξι παιδιών. Yeah, this is very worrying trend, not only in... Πολύ ανησυχητικό το φαινόμενο, όχι μόνο στην Ισπανία. Ε, τα μέλη μας ε, μας ενημερώνουν διαρκώς. Α, και το Equinet, ε, το δίκτυο των οργανισμών για την ισότητα σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο καταγγέλνουν αυτή τη διακριτική μεταχείριση λόγω εγκυμοσύνης. Πολύ δύσκολο είναι αυτό, διότι κανονικά απαγορεύεται. Και είναι όμως και καλυμμένη αυτή η πρακτική που την καποφλάρουνε οι εργοδότες Δηλαδή γίνεται μία προδιαλογή κατά τη διάρκεια της ε, πρόσληψης. Και παρότι απαγορεύεται για νόμο, ε, ε, επανεμφανίζεται αυτό το παλιό πρόβλημα πολύ δύσκολο να καταπολεμηθούν αυτά τα στερεότυπα που νομίζαμε ότι είχαν ξεπεραστεί. θα χρειαστεί όμως να επανέλθουμε και να συνεργαστούμε και με εργοδοτικές οργανώσεις για να υπάρξει ε, μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα περισσότερο αυτή τη στιγμή. Ευχαριστούμε κυρία Βυσνιεύσκα. Μια σύντομη ερώτηση και κατόπιν ο κύριος Ταραμπέλα. Μέχρι τις 7 παρα 20 έχουμε τους ε, διερμηνείς. Σας ζητώ να ε, συντομεύετε και στις ερωτήσεις και στις απαντήσεις. Κυρία Βυσνιεύσκα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Δεν θέλω να υπάρξει παρανόηση ότι ε, είναι κατά των γυναικών τα συνδικάτα στην Πολωνία ή δεν ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα, διότι δεν σταθεί αυτό. Νομίζω ότι αλλού έγινε το πρόβλημα. Η κυβέρνηση δεν εξάγει τον κατάλληλο διάλογο με, τις, ε, με τα συνδικάτα στην Πολωνία αυτά τα τελευταία 10-15 χρόνια. Δείτε το τι συνέβη με την μεταρρύθμιση του εξωτικού συστήματος και τη νέα ηλικία σε 67 για τους άντρες και για τις γυναίκες. Δείτε την ποιότητα ζωής ε, στις επαρχίες, στην Ήπεθρο. Βλέπετε πόσο χαμηλά είναι τα επίπεδα διαβίωσης, ε, οι διαγνωστικές πρακτικές, ε, η περίθαλψη. Είμαστε σε μαύρο κατάλογο στην Πολωνία. Θα ζητήσω από τους συναδελφούς να μην μιλούν εξ ονόματος ε, όλων των γυναικών, ε, διότι υπάρχουν και γυναίκες που πιστεύουν ότι είναι εξαιρετικά σημαντικά ε, τα παιδιά και η οικογένεια και διαφωνούμε με την κυρία Κοσλόφσκα. Ναι, εντάξει, τη της έδωσε, λέει η Προεδρεύουσα, ο κύριος Ταραμπέλα. Ευχαριστώ. Εγώ υπερψήφισα, αλλά μόνος μου είμαι ε, για την προηγούμενη παρέμβαση έκανε το αστείο κύριο Σταραμπέλα. Θα ήθελα να θυμίσω ότι είναι μια, ένας μόνιμος αγώνας η καταπολέμηση της βίας. Κάποια στιγμή ίσως συζητείται περισσότερο, άλλοτε λιγότερο, αλλά παρόλα αυτά. Ε, κάποια στιγμή Ξέρετε, το πιο συμβολικό εργαλείο του βουλευτή είναι η δήλωση ε, νομική. Νομικό βάρος δεν έχει, αλλά τέλος πάντων ε, ε, στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία στην αρχή είχαμε κάνει μια γραπτή δήλωση, είχα μαζέψει πάρα πολλές υπογραφές και ζητούσαμε τα επόμενα πέντε χρόνια, και ήταν το 2010, τα επόμενα πέντε χρόνια είχαμε ζητήσει να, να επιλεχθεί ένα έτος που θα ανακυρισόταν σε έτος καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών. Όχι ότι θα λύσουμε τα προβλήματα με αυτό το έτος. Ε, το ίδιο έγινε και με τη φτώχεια, δεν σημαίνει ότι λύθηκαν τα προβλήματα. Όχι, αλλά τέλος πάντων ε, είναι μια καλή προσπάθεια. Όλοι οι αρμόδιοι στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, στους εθνικούς φορείς, ε, στις οργανώσεις ε, μπόρεσαν να κάνουν μια ανταλλαγή απόψεων για ένα ζήτημα που σε ορισμένε χώρες είναι περισσότερο ταμπού. έτσι, συζήτησαν οι άνθρωποι, αναφέρθηκαν σε αυτό το ζήτημα και σίγουρα αυτό συνιστά πρόοδο για όσους υφίστανται το πρόβλημα. Για να ε, σημειώσει επιτυχία μια γραπτή δήλωση χρειάζονται 10 συνάδελφοι από τον ανώτερο δυνατό αριθμό ε, πολιτικών ομάδων και ε, από μεγάλο αριθμό χωρών κατά προτίμηση. Θα πρέπει να αποκτήσουμε νέα αντανακλαστικά. Ζητούμε αξιολόγηση αντικτύπου για τα φύλλα, για τις πολιτικές. Ε, μιλούσαν παραδείγματος χάρη για την εγγύηση για την νεολαία. Α, να, να ανοίξω και μια άλλη παρένθεση, θα την κλείσω σε λίγο. Έχω την εντύπωση ότι προς στιγμής είναι μια εξαγγελία και μόνο, διότι ακούω ότι σε κάποιες χώρες η ε, δημόσιοι φορείς ε, που θα το αναλάβουν, να δώσουν, ε, να προσφέρουν επιπρόσθετη μετεκπαίδευση ή ένα, μια πρακτική άσκηση ή μια θέση εργασίας έστω και προσωρινή για τους νέους, ε, για την πρώτη τους επαγγελματική εμπειρία ε, δεν έχουν τα απαιτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, λέει ο κύριος Γιούνκερ, ε, δεν θα δώσουμε παραπάνω λεφτά, Έξι Καλά είναι τα έξι δις, αλλά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν και λέει ότι δεν απορροφούνται τα κονδύλια. βέβαια δεν απορροφούνται, γιατί ε, λειτουργεί ως τροχοπέδι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει κάποιος να ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα και να ξέρουμε όλοι ότι φταίνε οι υπηρεσίε Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι οι εθνικοί φορεί που δεν απορροφούνται τα κονδύλια. Δεν πρέπει να υποτιμήσουμε ή να υποβαθμίσουμε αυτή την πολιτική, γιατί αλλιώ δεν θα έχει την αναμενόμενη επιτυχία. Ε, χρειάζεται ανάλυση ω προ την ισότητα των δύο φύλων με το κονδύλι που έχει προβλεφθεί για τα προγράμματα που ε, θα ε, δρομολογηθούν και προσοχή να μην στιγματιστεί η πολιτική λόγω ανισότητας ε, των δύο φύλων. Στην έκθεσή μου <clears throat> σε όλα τα επίπεδα θα ασχοληθούμε με αυτό το νέο αντανακλαστικό που πρέπει να ε, αναπτύξουμε και να εντάξουμε σε όλους τους νέους διαλόγους, σε όλες τις νέες ανταλλαγές ε, που θα κάνουμε. Εδώ. Ευχαριστώ. Θα σας θυμίσω το χρονοδιάγραμμα. Η παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης είναι 1-2 Δεκεμβρίου 2014, οι προθεσμίες υποβολής των υπολογιών 8 Δεκεμβρίου, έγκριση από την Επιτροπή μας ε, τον Ιανουάριο του 2015 και στην Ολομέλεια το Φεβρουάριο ελπίζουμε. Ευχαριστώ ε, την ομιλήτριά μα, σημείο 7, στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών με το 2015. Θα δώσω αμέσω το λόγο στην εισηγήτρια κυρία Μαρία Νόικλο να σα πω ότι 3 Σεπτεμβρίου του 2014 ε, οι συντονιστέ αποφάσισαν την υιοθέτηση μια έκθεση στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η μισότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το 2015. Το 2015 θα ξεκινήσει η Επιτροπή ε, την, νέα τη στρατηγική για την ισότητα των γυναικών και τι προτεραιότητε που θα δώσει ξελογώντας ε, την πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Η έκθεση πρωτοβουλία τη Επιτροπής Γυναικών θα αποτελέσει τη συμβολή του Κοινοβουλίου προ την Επιτροπή για τη διαμόρφωση νέα στρατηγική. Σήμερα θα έχουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την έκθεση ιδίες πρωτοβουλίε και κάποιες ιδέες για να σκεφτούμε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στην εισηγήτρια. Θυμηθείτε ότι μέχρι τις 7 παρα 20 έχουμε τους Γερμηνείς και άλλα θέματα επίσης στην ε, ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πω λίγα λόγια για κάποιες πρώτες σκέψεις ε, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών και κατόπιν θα με ενδιαφέρει να έχω σχετική συζήτηση μαζί σας. Ήδη αναφέρθηκε στην προηγούμενη έκθεση ότι 6-7 θέματα ε, έχουν ε, αποκρισταλωθεί, τα οποία θα πρέπει να υπάρχουν στην επόμενη έκθεση. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να ασχοληθούμε αποκλειστικά με τα θέματα αυτά. Είναι σημαντικό να παρουσιάσουμε τις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων θεμάτων, ότι για παράδειγμα η σεξουαλική βία έχει επιπτώσεις για τον χώρο εργασία των γυναικών, ότι αυτή εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση, ότι η οικονομική κατάσταση των γυναικών έχει συνέπειε για την υγεία τους κλπ. οποίο ε, διαμορφώνει πολιτική ισότητα πολύ σύντομα διαπιστώνει ότι δεν ε, μιλάμε για ε, ξεχωριστούς πυλώνες αλλά ότι, είναι για θέματα που, ότι μιλάμε για θέματα που είναι στεδεμένα μεταξύ τους. Θέλουμε λοιπόν να δείξουμε ότι ε, το θέμα που μας ενδιαφέρει δεν είναι τα μεμονωμένα θέματα, αλλά η σχέση μεταξύ τους. Οι γυναίκες ε, στην αγορά εργασίας είναι ένα κεντρικό θέμα, έχει να κάνει με την ισότητα ε, την μισθολογική, έχει να κάνει με τους παράγοντες που ρίχνουν στη φτώχεια τις γυναίκες και με τον συνδυασμό ιδιωτικού και επαγγελματικού βίου. Επίσης, ε, γυναίκες στην κρίση. Όταν δυσκολεύουν τα πράγματα εντός ενός ε, κράτους, ε, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερο ο ρόλος των γυναικών. Θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα στις γυναίκες και την υγεία. Αυτό δεν αναφέρθηκε στην προηγούμενη έκθεση ήταν ένα θέμα το οποίο ε, αναφερόταν παρεπιπτόντος. Είναι πολύ σημαντικό θέμα όμως, έχει να κάνει με την πρόσβαση στο σύστημα υγείας, έχει να κάνει με τις ε, ασφαλίσεις, έχει να κάνει όμως όλο και περισσότερο με το πώς διαμορφώνεται η πολιτική της υγείας και το πώς οι έρευνες, για παράδειγμα, επικεντρώνονται περισσότερο στο σώμα των ανδρών και όχι τόσο πολύ των γυναικών. Τέτοιες ε, διακρίσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την υποχρέωση να κοιτάξει και πέρα από τα όρια της. Δηλαδή όχι μόνο να διαμορφώσουμε πολιτική ισότητα για μας, αλλά να αναγνωρίσουμε ότι η πολιτική ισότητα στην Ευρώπη θα έχει συνέπειες και για την πολιτική ισότητα σε άλλα μέρη του κόσμου. Ε, στην στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής και της επίλυσης ε, συγκρούσεων ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το θέμα αυτό, διότι βλέπουμε ότι αυτά συχνά είναι εις βάρος των γυναικών. Σκέφτομαι, για παράδειγμα, ότι θα πρέπει να αναφέρουμε την αναπτυξιακή συνεργασία. Είναι σαφές ότι η έκθεση αυτή, λόγω του στενού χρονοδιαγράμματος, δεν μπορεί να συμπεριλάβει όλα τα θέματα. Θα πρέπει όμως να καθίσταται σαφές από την αρχή με ποια θέματα ασχολούμαστε και να προχωρήσουμε με κάποια από αυτά. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τη γνώμη σας για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. Donc, je cède la parole. Σας ευχαριστώ. Ποιοι θα ήθελαν τον λόγο. Γκάλ Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Σωστή είναι η προσέγγιση που έχει οθετήσει. Συμφωνώ και εγώ. Πως όλα τα ζητήματα είναι αλληλένδετα, κυρίως σε αυτό το τομέα. Δεν είναι νέο αυτό το ζήτημα, δεν το συζητούμε πρώτη φορά σήμερα σήμερα. Βλέπουμε πως ε, τα όσα συμβαίνουν σήμερα συνδέονται επίσης άμεσα με ε, τα, την προηγούμενη περίοδο στρατηγικού προγραμματισμού 2010 έως 2015. Θα χρειαστεί να ακολουθούμε συγκεκριμένους προσανατολισμούς για να καταρτήσουμε στρατηγική ε, ε, για να καταρτιστεί η στρατηγική χρειαζόμαστε και τις μεθόδους και τα εργαλεία όταν ε, μιλάμε για την για την αναπτυξιακή συνεργασία, για τις γυναίκες στην κρίση. Θα πρέπει να βρούμε κάθε φορά τα κατάλληλα εργαλεία. Περισσότερα είναι δε τα εκκρεμή ζητήματα από αυτά για τα οποία έχει βρεθεί μια ικανοποιητική λύση, κυρίως ως προς τα ζητήματα αγοράς εργασίας. Λένε και περισσότερες γυναίκες ε, μπαίνουν στην αγορά εργασίας, ε, ε, ανέρχονται σε ανώτερες διοικητικές θέσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει αυξηθεί και η επιρροή τους. Αφήστε που ένας μεγάλος αριθμός έχει αποκλειστεί από την αγορά εργασίας και ζει κάτω από το όριο φτώχειας. Ε, είναι σημαντικό να δούμε την επιδείνωση ε, στο επίπεδο φτώχειας κυρίως για τις ηλικιωμένες γυναίκες. Επίσης, θα χρειαστούμε κατάλληλους δείκτες για να καταμετρηθεί η πρόοδος ή η απουσία πρόοδου. Για το, την εγγύηση για την νεολαία ή για το ζήτημα του συνταξιοδοτικού χάσματος είναι δύσκολο να ξέρουμε σε τι αποβλέπουμε Πολύ δύσκολα μπορούμε να έχουμε ένα κοινό στόχο όταν έχουμε ε, ενισχύει 28 διαφορετικά συστήματα. Χρειαζόμαστε όμως απεραγκλήτως κοινούς στόχους Και να μην ξεχνάμε ότι η εξασφάλιση της ισότητας των δύο φύλων μπορεί να λειτουργήσει ως ε, κινητήριος δύναμη για την ε, ανάκαμψη της οικονομίας. Θα ήθελα να καλυφθούν όλα αυτά τα επιμέρους ζητήματα στη στρατηγική που θα προτείνουμε. Σίγουρα δεν είναι ρεαλιστικό να περιμένει κανείς να εξαλειφθούν τελείως τα χάσματα που υπάρχουν. Θα μπορούσαμε τουλάχιστον όμως να ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μια καλύτερη συνεργασία. Είναι υποχρέωση για μας, δεν είναι μόνο μια δυνατότητα που έχουμε, είναι υποχρέωση για μας να κάνουμε κάτι διότι οι γυναίκες περιμένουν αυτή τη στρατηγική για την περίοδο μετά το 2015. Έχουμε το πλαίσιο για κάποιο περιθώριο ελιγμών και παρότι όμως Είμαι καινούργιο μέλος στην Επιτροπή. Έχουν εντύπωση δεν έχουμε εξαντλήσει το διαθέσιμο προϋπολογισμό. Ας χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τις δυνατότητες που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας και μετά ας περάσουμε στο επόμενο επίπεδο. δηλαδή να μπαίνουμε στα χωράφια των κρατών μελών και στις δικές τους αρμοδιότητες. Ευχαριστώ. Ποιος άλλος θα ήθελε τον λόγο. Κύριε Βυσνιεύσκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, με χαρά μπορώ να σας πω ότι στη στρατηγική που προετοιμάσαμε δεν υπάρχει έμφαση στην πολιτική υγείας και περισσότερη υποστήριξη για τις γυναίκες ό,τι αφορά την προστασία της υγείας τους. Ιδίως στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Η Ευρώπη έχει μια κρίση δημοκρατική και να προωθήσετε την μητρότητα και να συμπεριληφθεί στην στρατηγική που ετοιμάζουμε. Μιλήσατε για τις ανισότητες προς τις γυναίκες. Αυτό ισχύει στην Πολωνία. Θέλω να σας θυμίσω ότι αυτό είναι εθνικό ζήτημα που αποφασίζεται σε εθνικό πλαίσιο. Ας προστατεύσουμε λοιπόν τις γυναίκες, αλλά ας τις υποστηρίξουμε, αλλά ας μην πάμε από τη μία άκρη στην άλλη. Ας μην παρεμβαίνουμε σε τομείς που δεν υπάγονται στη δική μας αρμοδιότητα. Ευχαριστώ. Άλλος. Κάποιοι από την Επιτροπή θέλουν το λόγο. Ξανά. Ευχαριστώ. Τέτοια ώρα που είναι, καλωσορίζω την ε, συζήτηση που ξεκινήσατε. Είναι σημαντικό θέμα για μας. Σε κρίσιμη στιγμή έρχεται συζητούμε το θέμα της ισότητας ε, εν ώψη της προετοιμασίας ε, της ατζέντα ε, για την Ένωση μετά την, το 2015 θα υπάρξει θα δώσουμε έτσι το πλαίσιο των μελλοντικών συζητήσεων πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία και με χαρά να συνεχίσουμε την συνεργασία στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπιόρκ. Προσβλέπω στην καλή συνεργασία με την εισηγήτρια ώστε να γίνει αυτή η έκθεση όσο γίνεται καλύτερη. Ε, όλα ακούστηκαν πολύ καλά, αλλά θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Ε, με ανησυχεί λίγο Κάποιοι θα θέλουν όλους τους λόγους διακρίσεων σε μια στρατηγική ε, για την ε, ισότητα. Θέλουμε μία στρατηγική ισότητα με φιλόδοξους ε, στόχους και να επιλέξουμε τους πιο σημαντικούς τομείς για μας και πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ως πρώτη παρατήρηση στην έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αν δεν θέλει κάποιος άλλος ε, τον λόγο, θα δώσω το λόγο στην ε, εισηγήτρια για τα συμπεράσματα. Ε, στο προσεχές διάστημα θα είναι ανοιχτή η πόρτα μου. Θα ήθελα πολύ να ακούσω οποιασδήποτε σκέψεις. αν κάνουμε ο καθένας από ένα μικρό βήμα, θα γίνει τελικά ένα μεγάλο βήμα. Ευχαριστώ. Να σας συμβήσω το, το χρονοδιάγραμμα. Το σχέδιο έκθεσης ε, θα υποβληθεί 20 Ιανουαρίου, προθεσμία υπολογιών 27 Ιανουαρίου, εξέταση των τροπολογιών 26 Φεβρουαρίου, έγκριση στην Επιτροπή Γυναικών 30-31 Μαρτίου του 2015 και στην Ολομέλεια τον Απρίλιο του 2015. Προχωρούμε τώρα στο σημείο 8. Ευρωπαϊκή Ένωση και Παγκόσμιο Πλαίσιο Ανάπτυξης με το 2015. Θα δώσω αμέσω του λόγου στην κυρία Μπιόρκ για να μας εξηγήσει στο λίγο χρόνο που έχουμε τι περί τίνος πρόκειται. Ίσως να έχουμε και λίγο χρόνο συζήτησης. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομη διότι έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Η έκθεση αυτή έχει επίσης πολύ στενό χρονοδιάγραμμα. Έχουμε εργαστεί πολύ γρήγορα ώστε να έχετε μπροστά σας ε, την το σχέδιο έκθεσης. Αν κατάλαβα σωστά, η Γραμματεία θα ανακοινώσει την ε, ε, ε, προθεσμία για τις τροπολογίες που είναι αυτή την Παρασκευή. Έχουμε λοιπόν πολύ λίγο χρόνο. Θα ήθελα όμως να τονίσω κάποια από τα πράγματα που έχουμε κάνει. Οι εργασίες έχουν βασιστεί στις εργασίες της Επιτροπής μας κατά τη διάρκεια της τελευταίας θητείας και αναφερόμαστε στους νέους στόχους μετά το 2015 και βλέπετε στα θέματα που τονίζουμε στο σχέδιο της έκθεσης ε, ότι θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένους στόχους στο νέο πλαίσιο που θα ισχύσει μετά το 2015 και πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εδώ μεγάλη υποχρέωση να πιέσει στις διεθνείς διαπραγματεύσεις και είναι σημαντικό ως Κοινοβούλιο να στείλουμε σαφές μήνυμα. Επίσης, στο σημείο 3, τονίζουμε κάποιους τομείς όπου είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει ισότητα σε διεθνές επίπεδο. Μιλάμε για την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, στην εκπαίδευση, στην καταπολέμηση της στόχιας, στην ενίσχυση της οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών, να καταπολεμούσουμε την βία εις βάρος των γυναικών και να ε, βελτιώσουμε την πρόσβαση των γυναικών ε, σε υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας. Έχω σκεφτεί κάποια θέματα τα οποία θα ήθελα να αποτελέσουν αντικείμενο τροπολογιών. Για παράδειγμα, να έχουμε ξεχωριστή παράγραφο σχετικά με την αναπαραγωγική υγεία και τα σεξουαλικά δικαιώματα. Να έχουμε μια παράγραφο για το διεθνέ εμπόριο διότι υπάρχουν και εδώ πτυχές ισότητας, ε, ενδεχομένως ε, μία παράγραφο για την καταπολέμηση της φτώχειας ε, από την πλευρά των γυναικών και επίσης ε, θέλουμε να αναφέρουμε τα ε, δικαιώματα των ε, ατόμων ΛΟΑΔ. Ξέρω ότι είναι πολύ στενό το χρονοδιάγραμμα, αλλά ελπίζω ότι θα μπορέσουμε μαζί να διαμορφώσουμε μια καλή έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Κυρία Ρενά, θέλει το λόγο. Γρήγορα, γρήγορα. Ευχαριστώ για όσα μας είπατε εντάχει που περιέχουν τις προτεραιότητες. Είναι σημαντικό νομίζω να δούμε το θέμα των ε, νέων των, των κοριτσιών. Ο στόχος, δεν μιλάμε για ανάπτυξη, ο στόχος των κοριτσιών είναι σημαντικός και για την εκπαίδευση αλλά και για τα σεξουαλικά και παραγωγικά δικαιώματα. Πάρα πολλές νέες κοπέλες αυτή τη στιγμή είναι θύματα ε, γάμων σε μικρή ηλικία, που σημαίνει εγκυμοσύνη σε μικρή ηλικία, που σημαίνει υψηλή θνησιμότητα, η κίνδυνος υψηλής θνησιμότητας για τις νέες κοπέλες. Άρα η ομάδα αυτή είναι σημαντική στο πλαίσιο της ανάπτυξης. Ή είπα κι άλλα, εκπαίδευση υγείας και βία, υγεία και βία να πρέπει να ανηλύονται και από την οπτική της ηλικίας ε, στις κοπέλες ε, σε ανάπτυξη. Ευχαριστώ. κάποιο άλλο Αν δεν υπάρχουν, να σας θυμίσω ότι η προθεσμία για την κατάθεση των απολογιών είναι 17 Οκτωβρίου 10 το πρωί. 6 Νοεμβρίου θα εξεταστούν και θα ψηφιστούν την ίδια μέρα εδώ. Και στις 11 Νοεμβρίου στην Επιτροπή ΝΤΕΒΕ. Στην Ολομέλεια θα δούμε πότε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και τους διερμηνείς που έμειναν μαζί μας. Καλό βράδυ.